Welcome to everybody. Please. Uh, Να σας καλωσορίσω. Καθίστε παρακαλώ. And we can start now. Θα ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και με τους συναδέλφους που φιλοξενούμε αυτή την πολύ σημαντική διακοινοβουλευτική συνεδρίαση. Ξεκινήσα στα αγγλικά, θα συνεχίσω στα ιταλικά φορέσετε λοιπόν τα ακουστικά σας. Χαίρομαι λοιπόν που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, στα δύο πάνελ που θα έχουμε και έχουμε και έχουμε εκπροσώπους από την Σλοβακική Προεδρία, τον κύριο Άντων Σκρέκο, ο οποίος είναι Γενικός ε, Διευθυντής ε, Οπτικοακουστικών Μέσων και το Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης ε, και Πολιτισμού από την Κομισιόν, την κυρία Μάρτιν Ράικερς. Έχουμε 31 μέλη από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση και έχουμε εδώ φυσικά και συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως μέλη της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Πολιτισμού και ε, θα σας τους παρουσιάσω φυσικά στη διάρκεια των εργασιών και ε, ε, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ. Ξέρω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει αυτή η συνεδρίαση σήμερα. Πριν περάσω στα Ιταλικά θα ήθελα να σας πω ότι Πρόκειται για τη δεύτερη διακοινοβουλευτική συνάντηση που διοργανώνουμε ως Επιτροπή Πολιτισμού. Ως πρόεδρος ε, μαζί με τις ε, ε, πολιτικές ομάδες στις Επιτροπής αποφασίσαμε να ξεκινήσει αυτή η σημαντική συνάντηση για να ακούσουμε και τις προτάσεις σας, να υπάρξει μία συζήτηση με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων ώστε να δημιουργήσουμε δεσμούς και να δημιουργήσουμε μαζί έναν ευρωπαϊκό χώρο πολιτισμού. Πέρσι αφιερώσαμε την διακοινοβουλευτική συνεδρίασή μας ε, στην παιδεία και στην νεολαία και φέτος, όπως γνωρίζετε, στον πολιτισμό και στη δημιουργικότητα εν γέννη, αλλά ε, επικεντρωνόμαστε στα θέματα αυτά. Τώρα θα περάσω στα Ιταλικά. Φαντάζομαι ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα με τα ακουστικά. Μπορείτε να βρείτε το κανάλι των γλωσσών που σας ενδιαφέρουν ώστε να νιώθετε εσά στο σπίτι σας και να ακούτε τη γλώσσα σας. Ωραία, θα περάσω τώρα στα Ιταλικά, να σας πω απλώς ότι σας ευχαριστώ πολύ και γιατί οι περισσότεροι από εσά απαντήσατε με πολύ ενδιαφέρον τρόπο στο ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε, το οποίο εστίαζε σε τέσσερα σημεία στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών, και στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα στις χώρες σας. Ε, τι πολιτικές εφαρμόζονται στον τομέα αυτό, τι δράσεις έχουν ξεκινήσει προκειμένου να συμμετέχουν και οι πολίτες ε, στην πολιτιστική δράση, που είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν, και τι άλλο ε, ζητάτε να αναπτύξει η Ευρώπη και κυρίως ποιες είναι οι προκλήσεις για σας στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό και αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζουμε να έχουμε πλέον ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, αν και ακόμα βρίσκεται στα σπάργανα, και φυσικά ε, δεν έχουμε πλήρη επικουρικότητα ε, όπως έχουμε στον πολιτισμό. Η δημιουργικότητα όμως έδωσε όθηση και μέσω των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκθέσεών μας, αλλά και μέσω των συμπερασμάτων των διαφόρων συμβουλίων υπουργών, ε, από το θεματολόγιο για το 2015-2017 το οποίο εγκρίθηκε στην Ιταλική Προεδρία. Ε, στη συνέχεια δόθηκε ε, μια πολύ μεγάλη όθηση από την επόμενη Προεδρία στην δημιουργικότητα και στον πολιτισμό και αυτή τη στιγμή ε, προχωρούν ιδιαίτερα αυτά τα θέματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια στρατηγική καμπή για να δώσουμε την κατάλληλη όθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και με τη βοήθεια των κρατών μελών. Από τα διάφορα αιτήματα και τις προτάσεις σας μου φαίνεται ότι ανακύπτει η ανάγκη να υπάρχει ένα σαφέστερο νομικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να έχουμε τα στοιχεία της ε, δημιουργικότητας και του πολιτισμού στην Ευρώπη. Ε, υπάρχουν επίσης αιτήματα για να δώσουμε όθηση για την καινοτομία και ε, ως ε, άξονας ανάπτυξης ε, και ως προοπτική κοινωνικής ένταξης, ε, τα θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, και νέα μοντέλα διαχείρισης, σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα για παράδειγμα που είναι ένα από τα θέματα τα οποία προωθήσαμε αυτά τα χρόνια και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να τα προσαρμόσουμε και στις νέες ψηφιακές προκλήσεις ε, για τις συγκεκριμένε ανάγκες του πολιτισμού, των δικαιωμάτων του δημιουργού κλπ. που είναι θέματα που και αυτά συζητούμε μέσω οδηγιών στα πλαίσια της στρατηγικής ε, για το ψηφιακό ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Και βεβαίως ε, διαπίστωσα με ευχαρίστηση, με ως μόνιμη ε, εισηγήτρια για την ε, δημιουργική Ευρώπη ότι κάποιοι από εσά ζήτησαν πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση για αυτό το πολιτέ πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει υποπρογράμματα το Μέντια και το Κουλτούρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή και στο οποίο έχουν δοθεί ένα δισεκατομμύριο 400 ε, εκατομμύρια ευρώ για την τετραετία αυτή και πραγματικά εκφράσατε την επιθυμία να ξεκινήσει το νέο ευρωπαϊκό μέσο για την εγγύηση ε, για τις ε, ε, τράπεζες οι οποίες θέλουν να προσφέρουν δανειοδότηση. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ιδιαίτερα τα θέματα αυτά και να υπάρξει και κατάλληλη πολιτική βούληση. Χωρίς κατάλληλες επενδύσεις και χωρίς κεντρικό ρόλο για τον πολιτισμό, ελοχεύει ο κίνδυνος να μην υπάρχει μέλλον για την Ευρώπη, αλλά να μην υπάρχει και βιώσιμη ανάπτυξη. Πάντα αναφερόμαστε σε η βιώσιμη, ευφυή ε, ανάπτυξη που περιλαμβάνει τις πάντες. Πολύ δύσκολα μπορούμε να το πετύχουμε αυτό χωρίς να έχουμε και προώθηση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών στοιχείων. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω, εδώ και πολύ καιρό λέμε ότι ο πολιτισμός είναι ο τέταρτος πυλώνας της βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Εάν δεν γνωρίζουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, αν δεν υπάρχει πρόσβαση στον πολιτισμό και αν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκφράσουμε τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά μας ένστικτα, δεν ανανεωνόμαστε. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε γιατί θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα αυτά και στα κράτη-μέλη. Ξέρετε ότι οι δύο πυλώνες της Δημιουργικής Ευρώπης περιλαμβάνονται στη συνθήκη, η προώθηση της ε, πολιτιστικής ε, και γλωσσικής ποικιλομορφίας αφενός και αφετέρου η προστασία και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ε, στοιχεία τα οποία λοιπόν ε, μας οδηγούν στο να μην θεωρούμε κρατική ενίσχυση της ενισχύσεις για τα θέματα αυτά, αλλά ως ένας τρόπος για να εγγυηθούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, τον πολιτιστικό μας πλούτο που είναι η πραγματική αξία της Ευρώπης στον κόσμο. Βεβαίως πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει περισσότερο στο επίκεντρο του θεματολογίου της τα θέματα αυτά. Στην αρχή εμείς δεν ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι διότι δεν υπήρχε κάποια προτεραιότητα μεταξύ των 10 προτεραιοτήτων που παρουσίασε ο Πρόεδρος κύριος Γιούνκερ για τον πολιτισμό και πιστεύω και βλέπω και τους αδέλφους εδώ που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό ότι εμείς κάναμε αυτό που μας αναλογεί και θα σας πω πολύ γρήγορα προς ποια κατεύθυνση διότι υπάρχουν περαιτέρω προκλήσεις οι οποίες ε, ε, σημαίνουν ότι πρέπει σε αυτή την εγκάρσια διάσταση των ε, ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών να προσδώσουμε μεγαλύτερη αξία όπως για παράδειγμα τα τραγικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη ε, και στην Μεσόγειο, τα κατεπίγους ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται, αλλά και πολιτιστικές συγκρούσεις. Εάν δεν δημιουργήσουμε γέφυρες και δεν υψώσουμε τύχη, εάν δεν έχουμε διάλογο και δεν έχουμε ε, κλειστή συμπεριφορά, ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και ο πολιτισμός μπορεί να τα προσφέρει αυτά. Από τη μια μεριά λοιπόν Υπάρχει αυτό το οποίο υπερασπιστήκαμε με στένος, ε, ξεκινώντας από την πολύ σημαντική έκθεση του κυρίου Διακόνου. Σήμερα συζητήσαμε την περιβόητη απόφαση που ελήφθη επιτέλους ε, το 2018 να είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα αποτελέσει μια ευκαιρία να δούμε την ευρωπαϊκή διάσταση της άειλης και ηλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα άλλο στοιχείο σε αυτή τη λογική είναι αυτό το οποίο χαιρετήσαμε με πολύ θετικό τρόπο και το οποίο ζητήσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το οποίο εγγενίασε η κυρία Μογκερίνη με τον ε, Επίτροπο Αναβράτση και τον Επίτροπο Χάν, ο οποίο είναι υπεύθυνο για την πολιτική γειτονία και μαζί με την ανακοίνωση για την Ευρώπη ω πολύ σημαντικό στοιχείο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το διάλογο, για αυτό γιατί είναι δύσκολο, πρέπει να υπάρχει και νέα πολιτιστική διπλωματία. Εμεί ε, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε την ε, προσέγγιση που είχαμε ε, στο παρελθόν που ακολουθούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ είμαι η συγγήτρια μαζί με τον συνάδελφο Μπρόκ, ο οποίος εκπροσωπεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτό για να σας πω ότι προσπαθούμε να ασχοληθούμε με οριζόντιο τρόπο με τα θέματα αυτά. Ε, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό το οποίο θα συζητήσετε εσείς, ε, τα εκπαιδευτικά πολιτιστικά ζητήματα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι πολλά υποσχόμενο, μπορεί να δημιουργήσει απασχόληση, κυρίως για τους νέους, καινοτομία και πάλι. Αν μου επιτρέπετε, καινοτομία δεν είναι μόνο τεχνολογική, υπάρχει πολιτιστική, κοινωνική καινοτομία και καινοτομία για όλους τομείς που μπορούμε να προωθήσουμε. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ε, γι' αυτό, διότι υπάρχει έκθεση του ε, συναδέλφου Μόργανο μαζί με τον συνάδελφο Έλερ από την Επιτροπή Βιομηχανίας για τις ε, προκλήσεις αυτές. Λέγεται ότι αυτή η καινοτομία πρέπει να είναι το 5 με το 8% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και θα μας βοηθήσει περισσότερο. Αυτό θα τα συζητήσετε και στο πάνελ. Μας ενδιαφέρουν επίσης οι δεξιότητες. Ε, αναφέρθηκε ε, και παρουσιάστηκε το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τις ε, δεξιότητες. Εμείς ζητούμε και συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Απασχόλησης για το θέμα τα αυτά, διότι θεωρούμε ότι οι αρμοδιότητες και οι δεξιότητες στην κατάρτιση, στον πολιτισμό και στην παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να βρουν το χώρο τους. Υπάρχει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη στην Ευρώπη για τα θέματα αυτά. Ένα άλλο θέμα είναι να μπορέσουμε να αντλήσουμε διδάγματα από τις θετικές εμπειρίες που είχαμε αυτά τα χρόνια, παραδείγματος χάρη οι πολιτιστικές πρωτεύουσε. Είμαστε στα 30 χρόνια αυτής της εμπειρίας, μια εμπειρία που ε, θα ήθελα αν καταφέρουμε μέχρι το Δεκέμβριο, αν δεν τα καταφέρουμε μέχρι το Δεκέμβριο αργότερα, θα το αποφασίσουμε με τους αδέλφους από την Επιτροπή Πολιτισμού, θα θέλαμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά για τις πολιτιστικές πρωτεύουσε, διότι στα 30 χρόνια υπάρχουν ε, ομάδες οι οποίες ξανασκέφτηκαν τις πόλεις, ε, προσπάθησαν να έχουν νέα κοινωνική ένταξη και νέα ηθαγένεια για να νιώθει κανείς πολίτης μέσα στην πόλη του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσουμε και πρέπει να την αξιοποιήσουμε καταλήλως. Επίσης, ε, πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι ε, σήμερα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, το βλέπουμε από τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου, με την κρίση μειώθηκαν ε, τα κονδύλια για τον πολιτισμό και την παιδεία, τεράστιες περικοπές, κυρίως ε, στη χώρα μου και επιτέλους σήμερα μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα. Ήταν μια ζωφερή και μακρά περίοδος και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στον πολιτισμό πλέον και στην παιδεία, διότι κατέρευσαν ε, και τα πολιτιστικά καταναλωτικά στοιχεία σε κάποιες περιπτώσεις. Πρέπει να υπάρχει δικαίωμα στον πολιτισμό και στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ε, κοινωνική ισότητα και σε αυτό το τομέα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι επί του θέματος αυτού ε, δέχτηκε την ευαισθησία που έχουμε ε, υπάρχουν δύο προσκλήσεις υποβολής προσφορών, η μία για τη μετεγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων μέσω της Δημιουργικής Ευρώπης και μία άλλη μέσω του Εράσμους. Πρόκειται για πρακτικές οι οποίες πρέπει να γίνουν πολιτικές, διότι αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να επενθυμίσω, διότι σας παρουσίασα μία πανευρωμική εικόνα για τα πάντα, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα. Αυτή τη στιγμή με δύο συναδέλφου που είναι συνεισηγήτριε, την κυρία Φερχάιεν και την κυρία Καμερέβερντ, ε, συζητούμε μια πολύ σημαντική οδηγία, την οδηγία για τι οπτικοακουστικέ υπηρεσίε και εδώ πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εξισορρόπηση των ε, δικαιωμάτων ε, και του δικτύου και της προστασίας ε, διαφόρων σημαντικών στοιχείων, προστασίας ανηλίκων και το καθεξής, αλλά και της ιδιαιτερότητας της δημιουργικότητας και των δημιουργών και αυτό ισχύει και για την οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα που θα συζητήσουμε εντός ολίγου μαζί με άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερους. Ζητώ συγγνώμη που τα λίγο τόσο γρήγορα, αλλά προσπάθησα λίγο να σας ενημερώσω για το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε και να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα, διότι πιστεύω ότι τελικά τα θεματολόγια μας μοιάζουν περισσότερο από όσο πιστεύαμε. Ε, για καιρό φαινόταν να ζούμε σε διαφορετικούς πλανήτες, αλλά ελπίζω ότι πλέον η Ευρώπη, που σε πολλά στοιχεία δεν δείχνει και την καλύτερη πλευρά της αυτή τη στιγμή και τη μεγαλύτερη ελληνική της, ελπίζω λοιπόν μέσω του πολιτισμού, μέσω της βοήθειας όλων μας, να μπορέσει να ξαναβρει την ταυτότητά της και κυρίως ε, την ταυτότητα του πολιτισμού, που είναι ταυτότητα διαλόγου, ε, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο, καταρχάς της Σλοβακική Προεδρία. Έχουμε τον κύριο Άντων Σκρέκο, τον οποίο σας παρουσίασα προλίγου. Ε, μπορείτε να λάβετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εξ ονόματος της Σλοβακικής Προεδρίας. Παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή για μένα που μπορώ να σας απευθύνω το λόγο σήμερα και εκ μέρους του Υπουργού Πολιτισμού της Σλοβακίας έχω την ευκαιρία να κάνω την εναρκτήρια ομιλία σήμερα στη συζήτηση για τον πολιτισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου, εκπροσωπώντας τη Σλοβακική Προεδρία, να μιλήσω σλοβακικά. Και πιστεύω ότι θα κινηθώ και εγώ στο ίδια γραμμή, όπως και η κυρία Πρόεδρό σας, σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και τη σημασία του για τη δημιουργικότητα και για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε συνειδητοποίηση των θεμάτων του πολιτισμού στην εκπαίδευση και στο πόσο ο πολιτισμός συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη ο πολιτισμός είναι και το έδαφος που μπορούμε να καλλιεργήσουμε την δημιουργικότητα και την ε, βιομηχανία της δημιουργίας. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να έχουμε νέο κεκτημένο, να έχουμε απαντήσεις στις νέες οικονομικές και κοινωνικές παγκόσμιες προκλήσεις, πάντοτε με γνώμονα την καινοτομία. Η δημιουργική οικονομία είναι πηγή ιδεών, είναι πηγή και θέσεων απασχόλησης συνάμα. Οι δημιουργικές βιομηχανίες, οι κλάδοι δημιουργικοί της οικονομίας δημιουργούν και θέσεις απασχόλησης και αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο, έχει συζητηθεί επανειλημμένος, παραμένει όμως επίκαιρο και θεωρούμε ότι είναι κοινή μας πραγματικότητα. Μιλούμε για διαφοροποίηση των κλάδων των εθνικών οικονομιών και της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας στο σύνολό τους στο σύνολό της. Όλα αυτά δείχνουν πόσο είναι απαραίτητο να αλλάξουμε άποψη για την παραδοσιακή οικονομία, στο πλαίσιο δηλαδή της δημιουργικότητας. Πρέπει να δούμε όλους τους κρίκους αυτής της αλυσίδας έτσι ώστε να έχουμε δημιουργική παραγωγή, παραγωγή δημιουργικών προϊόντων, δημιουργική παρουσίαση, εκ νέου παρουσίαση ε, εξαγωγών, ε, αρχιοθέτησης και αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μία από τις υποσχόμενες πηγές ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πολιτισμός και αυτό έχει αποδειχθεί όλο και περισσότερο μεγαλύτερη μερίδα του ΑΕΠ καταλαμβάνει. Ε, βοηθά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και έτσι να συμβάλλουμε στη κοινωνική συνοχή και με αυτόν τον τρόπο καταπολεμούμε την οικονομική ύφεση. Η βιομηχανία της δημιουργίας και του πολιτισμού δραστηριοποιείται σε διάφορα πεδία καινοτομίας. και έχει αντίκτυπο θετικό όχι μόνο στις τέχνες και στον πολιτισμό, αλλά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας που απασχολούνται εκεί. Δική μας δουλειά είναι να έχουμε το σταθερό πλαίσιο, το ζωτικό πλαίσιο, για να επιτρέψουμε τη δημιουργία καινοτομία στον πολιτισμό, και έτσι η δημιουργικότητα και οι σχετικές δράσεις θα αποτελήσουν μέρος όχι μόνο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων αλλά και των ε, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από την πλευρά την οπτική γωνία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού και μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Μπορούμε να έχουμε μεγάλες συνέργειες. Μιλούμε για την παραγωγή, τη δημιουργία και τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών και αυτό θα ενισχύσει την ανάπτυξη. Υπάρχει και το διανοητικό κεφάλαιο, το πνευματικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να ενισχύσουμε. Δεν περιορίζονται όλα αυτά στις τέχνες. Βεβαίως υπάρχει περιθώριο δημιουργίας εισοδήματος από το εμπόριο αυτών των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αυξάνεται η οικονομική αξία και ενισχύεται η αγορά. Βασική στόχη για τη δημόσια πολιτική είναι ο πολιτισμός και η βιομηχανία της δημιουργίας να έχουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο ε, στη στο, δημιουργία του εθνικού ΑΕΠ και να έχουμε ένα σταθερό και συστηματικό πλαίσιο για να στηρίξουμε την καινοτομία στο πεδίο του πολιτισμού. Ε, θέλουμε να ενισχύσουμε τις συνέργειες με δημόσιες και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης, να διευκολύνουμε αυτές τις δυνατότητες έτσι ώστε κάθε δημιουργική συνεισφορά να αποτελέσει μέρος επιχειρηματικής δραστηριότητας και έτσι να συγχρονίσουμε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Θα έχουμε ένα αποτελεσματικό οικοσύστημα και θα έχουμε ε, άτομα και μονάδες που θα είναι πολύ πιο δραστηρία και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κινητοποιούνται έτσι οι ανθρώπινοι πόροι που αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες και θα πρέπει εμείς να ενισχύσουμε την εκπαίδευση, τα συστήματα εκπαίδευσης από την πιο μικρή ηλικία μέχρι και τη μεγαλύτερη έτσι ώστε να καλλιεργήσουμε ένα πνεύμα δημιουργικότητας και καινοτομίας θα πρέπει όλα αυτά να είναι μέρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ε, η δημιουργικότητα έτσι ώστε να αποκτήσει και αξία στην αγορά και να μπορεί να τύχει στήριξης και επένδυσης από τον ιδιωτικό τομέα. Και θα πρέπει να ειστηρίξουμε οικονομικά όλες αυτές τις δραστηριότητες, κυρίως όταν τις αναλαμβάνουν πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως προς τη βιομηχανία του πολιτισμού, ένα από τα βασικά είναι ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την αποτελεσματική προστασία και εφαρμογή της νομοθεσίας για θέματα πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας, που άλλωστε είναι και η ραχοκοκαλιά ε, του συστήματος. Σήμερα Έχουμε διάφορες αγωγές με τις οποίες ασχολούμαστε, έχουμε διάφορους φακέλους με τους, οποίου, τους οποίους μάλλον εξετάζουμε. Έχουμε το πρώτο πακέτο μεταρρυθμίσεων στο θέμα του copyright και τώρα έχουμε το δεύτερο πακέτο έτσι ώστε η προστασία του copyright να είναι πιο αποτελεσματική. Βεβαίως δεν περιοριζόμαστε εκεί, θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τη δημιουργία περιεχομένου για να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα σε όσο το πιο ευρύ πολιτιστικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Συμπερασματικά λοιπόν από τη δική μου πλευρά Θέλω να πω ότι ο κοινό παρανομαστής όλων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην βιομηχανία της δημιουργίας και του πολιτισμού είναι πώς θα ενθαρρύνουμε μια δημιουργική παραγωγή χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία, εστιάζοντας την προσοχή μας στη θεώρηση της ευρωπαϊκής οικονομίας ως αναπόσπαστο τμήμα των εθνικών, των εκάστοτε εθνικών οικονομιών. Ο πολιτισμός και η κουλτούρα δεν έχει να κάνει μόνο με την ταυτότητα, αλλά μπορεί να συνδεθεί και μάλιστα άρρηκτα με την ευμερία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ναι. πολύ για την εισαγωγή αυτή. Πολύ συγκεκριμένη, με πολύ σαφή στοιχεία. Ε, βασιζόμαστε στη Σλοβακική Προεδρία για δύο στοιχεία. Πρώτον, για να συντονιστείτε με τα όσα είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ, ότι δημιουργεί είναι τα κοσμήματα της κορώνας μας και θέλουν να θεωρούνται ως τέτοιοι. Ε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και δέσμευση από πλευρά Συμβουλίου, ώστε να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση και για την ε, Δημιουργική Ευρώπη και μια ad hoc χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς που αυτή τη στιγμή ε, σύμφωνα με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα επιβαρύνει τον προπολογισμό τη Δημιουργική Ευρώπη, που είναι πενιχρό ήδη. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει η συμφωνία του Συμβουλίου για να ξεπεράσουμε αυτέ τι δυσκολίε. Ευχαριστώ για τη διαθεσιμότητά σα και για τα όσα είπατε. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στη Μαρτίν Ράιχτερ, ε, η Γενική Διευθύντρια Παιδεία και Πολιτισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, είναι εξαιρετική τιμή για μένα που έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Η πρόεδρος μας, η κυρία Κώστα, κάλυψε ένα πολύ ευρύ πεδίο θεματικών ενωτήτων και δεν θέλω να τα επαναλάβω γιατί το έκανε πολύ καλύτερα από εμένα. Θέλω ωστόσο να σταθώ σε δύο-τρία στοιχεία. Όπως το είπε και η κυρία Πρόεδρος, πιστεύω ότι φέτο είναι ένα, ε, ένα σημείο καμπής στην ε, ε, επίσημη αφήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα λόγια του Προέδρου Γιούνκερ, ο οποίος είπε ότι οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες είναι τα ε, κοσμήματα του στέματος. Είναι μια έκφραση εξαιρετικά όμορφη, την οποία ε, θεωρούμε όλοι απολύτω έγκυρη, έγκυρη και επίκαιρη, ειδικότερα αν λάβουμε υπόψη μα το πόσα λίγα έχουν γίνει για την κουλτούρα και τον πολιτισμό τα τελευταία χρόνια. Αλλάζει η πολιτική λοιπόν τη Ένωση σε αυτό το πεδίο ε, φέτος και είναι θεμελιώδε αυτό, γιατί αν θέλουμε να απευθυνθούμε πραγματικά στι καρδιέ των Ευρωπαίων πολιτών, ε, θα πρέπει να μιλήσουμε με διαφορετικά λόγια και να μην επαναλαμβάνουμε συνέχεια ε, τα του ελλείμματος ή του εκάτα εκάστοτε οικονομικά στοιχεία, τα οποία ναι μεν είναι απαραίτητα, αλλά εν πάση περιπτώσει δύσκολα κάνουν τις ψυχές των Ευρωπαίων πολιτών να δονούνται. Σε κάθε περίπτωση όταν ανάλαβα τα καθήκοντά μου και ε, πρέπει να σας πω ότι δεν φανταζόμουν ότι θα είχαμε επιτυχία. Ε, σήμερα όμως είμαι η Γενική Διευθύντρια, η πιο ευτυχισμένη Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι είμαι επικεφαλής του προγράμματος Εράσμους, που είναι και το καλύτερο και το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διότι αυτά που γίνονται στο χώρο μας τα τελευταία, ε, τον τελευταίο καιρό είναι εξαιρετικά σημαντικά. Να ε, σταθώ λοιπόν σε αυτά που είπε η Πρόεδρος ε, σε ένα ή δύο σημεία και να πω το εξής. Ε, κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η κουλτούρα και ο πολιτισμός δεν τα βλέπουμε ξεχωριστά από τον υπόλοιπο κόσμο. Θεωρούμε ότι αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος του όλου. Και η έκθεση που έχει, έχουν, συνταχθεί, έχει, έχουν συντάξει τα μέλη σας ε, για τις βιομηχανίες της δημιουργίας δείχνουν ότι μπορούμε να ε, συνδέσουμε την κουλτούρα, τον πολιτισμό με τη δημιουργία. Δηλαδή δεν θα είναι η κουλτούρα από τη μία μεριά και η οικονομία από την άλλη. Είναι δύο κόσμοι τους οποίους έχουμε φέρει σε αντιπαλότητα και αντιπαράθεση για πάρα πολλά χρόνια και κακώς. Οι δημιουργοί πρέπει να έχουν τα προστοζήν για να είναι σε θέση να δημιουργήσουν και ο κόσμος της οικονομίας ο κόσμος γενικότερα χρειάζεται ε, τους δημιουργούς γιατί του προσφέρουν μια νέα θεώρηση των πραγμάτων με όχι αμυγός στεγνά και στενά ε, οικονομικά κριτήρια. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν θερμά για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής. Η Σίλβια απαρίθμησε τις δράσεις που δρομολογούνται, δεν θα τις επαναλάβω. Είμαι εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι έτσι θα κερδίσουμε αρκετό χρόνο. Δύο λόγια να πω για τη δέσμη ε, μέτρων Digital Agenda, ψηφιακή ατζέντα. Μετά τα κοσμήματα του στέματος που είναι πραγματικά σημαντικά, ε, το ε, πιο σημαντικό είναι οι δημιουργοί μας να έχουν τη δίκαιη ανταμοιβή. Και δεν έχουμε βρει ακόμα το καλύτερο σύστημα γι' αυτό, να αμείβονται δίκαια. Και όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, ε, είδαμε τελικά ότι δεν ήταν και η καλύτερη λύση να λάβουμε υπόψη τις πλατφόρμες. Ο Επίτροπος Ναβράτσιτς και εγώ ο ίδιος δώσαμε τεράστια μάχη για να ανοίξουν αυτές οι πλατφόρμες και να μην θεωρούνται μόνο ως χώρια ανταλλαγής απόψεων, αλλά να κομίσουν πραγματική προστιθέμενη αξία. Επομένως, δεν είναι αυτό που θέλετε να δείτε, δεν είναι αυτό που είναι το ευκταίο, όμως εδώ που είμαστε, είμαστε πολύ καλύτερα από εκεί που ξεκινήσαμε και θα πρέπει να καλύψουμε και την ε, υπόλοιπη απόσταση. Ο κόσμος της μουσικής είναι αυτός που επλήγει περισσότερο με τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή και είναι και αυτός που άλλαξε περισσότερο. Με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της δικής σας Επιτροπής κυρία Κώστα συνεχίζουμε θελήσαμε να συνεχίσουμε την πιλωτική δράση, δεν τα καταφέραμε, αλλά ας μην χάσουμε κάθε ελπίδα. Θα πρέπει να ε, καταλήξουμε ε, σε αυτό το συμπέρασμα. Υπάρχουν πλατφόρμες που μπορούμε νόμιμα να ε, φορτώσουμε ή να κατεβάσουμε μουσικό περιεχόμενο και αυτό να είναι παράδειγμα που θα χρησιμεύσει και σε άλλα πεδία του πολιτισμού. Ας μην απογοητευόμαστε λοιπόν. Δεν θα επαναλάβω ό,τι είπατε όπως είπα. Είμαι στη διάθεσή σας και είμαι έτοιμη να σας ακούσω και να απαντήσω σε κάθε ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις επισημάνσεις σας. Όντως υπάρχουν κάποια θέματα από των οποίων πρέπει να ενισχύσουμε ε, κάποια κοινά προγράμματα ε, ή κάποιες δράσεις οι οποίες ενισχύουν και το συντονισμό μεταξύ πολιτισμού και οικονομίας και φυσικά ε, δεν πρέπει να διατηρήσουμε μόνο τον πολιτιστικό χαρακτήρα αλλά πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το στοιχείο αυτό να δούμε λίγο κάποια οργανωτικά θέματα. Έχουμε δύο θεματικές ε, ενότητες. Ε, η πρώτη ε, είναι διαιρεμένη σε δύο πάνελ, γιατί ήταν αρκετοί οι βουλευτέ που θέλουν να παρέμβουν. Η πρώτη αφορά τι στρατηγικέ για την προώθηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Ο κύριος Βανσάν Λεπάζ θα κάνει την εισαγωγή. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ από την ε, Δημιουργική Βαλονία. Παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα σε πέντε λεπτά. Υπάρχει το πρόγραμμα πλαίσιο για την ε, ε, δημιουργικότητα στην Βαλονία. Θα μιλήσετε από τη θέση σα. Ε, δεν χρειάζεται να αλλάζουμε συνέχεια θέσει γιατί θα καθυστερήσουμε. Μετά θα ακούσουμε τρει βουλευτέ. τον κύριο Πατρίκ Βλός, ε, πρόεδρο τη Επιτροπή ε, Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων τη Γαλλική Εθνοσυνέλευσης, για πέντε λεπτά και πάλι. Μία ε, ιδιαίτερη προσωπικότητα για μας, την Εντίτε Στρέλα που διετέλεσε και ευρωβουλευτής, την ευχαριστούμε. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού για την συνέλευση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και στη συνέχεια ο κύριος Λουίτζι Μόργανο, ε, ο οποίος όπως υπενθυμίσαμε είναι εισηγητής της ε, έκθεσης για την ε, συνεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους να παραμείνουν σε αυτά τα πέντε λεπτά. Δυστυχώς αλλιώς θα υπο υποχρεωθώ να χρησιμοποιήσω αυτό το σφυράκι που δεν μου αρέσει να το χρησιμοποιήσω. Ε, χρησιμοποιώ, θα το χρησιμοποιήσω, ε, όχι επάνω σας βεβαίως, εδώ στο βήμα, ε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλους. Να δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στον κύριο Λεπάζ, στη συνέχεια, μετά από αυτές τις παρεμβάσεις, εάν υπάρχει ε, ε διάθεση μπορεί να παρέμβουν ελεύθερα όποιοι το επιθυμούν και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Ε, έχουμε τρία πάνελ, οπότε θα πρέπει να τηρήσουμε λίγο τους χρόνους. Παρακαλώ, ο κύριος Λεπάζ. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, Εγώ λοιπόν θα πρέπει να δώσω το παράδειγμα και θα είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω να ε, ανταποκριθώ στην πρόκληση. Με δύο λόγια λοιπόν, το Creative Valonia είναι πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2010 για να υποστηρίξει την ε, διάδοση της δημιουργικότητας στην οικονομία και στην ε, κοινωνία αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό θεωρήθηκε υποδειγματικό. Ε, δεν ε, θα σταθώ στα διάφορα στοιχεία τα οποία φαντάζομαι ότι τα έχετε μεταξύ των εγγράφων σα ε, για τα διάφορα αποτελέσματα τα οποία είχαμε τα πρώτα χρόνια Εκτέλεση αυτού του προγράμματο. Αυτό το οποίο έχει σημασία να αντιληφθούμε είναι ότι δεν ε, πρέπει να υποστηρίξουμε μόνο τη δημιουργική βιομηχανία, αλλά μπορεί να αποτελήσουν και μοντέλα, ε, ε, πηγέ υβριδικών μοντέλων και έμπνευση για του συγκεκριμένου αυτού τομεί. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του προγράμματο και θα σα πω αμέσω κάποια από τα αποτελέσματα για να μην χάσουμε χρόνο. Βλέπετε λοιπόν ότι τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα τα οποία αφορούν ε, κόσμο τον οποίο καταρτήσαμε, ευαισθητοποίησαμε, προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία διατέθηκαν στην αγορά και νεοφυείς υπηρεσίες, startups, οι οποίες, ε, ε, επιχειρήσεις οι οποίες υποστηρίξαμε. Πρόκειται λοιπόν κυρίως οικονομική, για οικονομική στήριξη σε πρώτη φάση. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να το τονίσουμε ε, κάτι το οποίο προώθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρήθηκε υποδειγματικό λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ε, στο European Creative District ε, που ξεκίνησε η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της δημιουργικότητας και την καινοτομία. Αν θυμάμαι καλά ήταν μια χρηματοδότηση η οποία συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για προπαρασκευαστικές δράσεις ε, για τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και χάρη σε αυτή τη χρηματοδότηση μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν αυτό το ε, πάρα πολύ σημαντικό ε, σήμα του European Creative District. Ε, επιλέγησαν δύο, η Τοσκάνη και η Βαλονία, επομένως ήταν μεγάλη τιμή για μας. Το πρόγραμμα αυτό μας επέτρεψε να δούμε κάποιες νέες προσεγγίσεις, ε, διάφορες πιλωτικές δράσεις, τις οποίες θα σταθώ στη συνέχεια και θα μας, μας επέτρεψε επίσης να ε, δούμε και ένα διεθνές πλαίσιο και με την Τοσκάνη, αλλά και με άλλες ε, περιοχές και χώρες της Ευρώπης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την Δημιουργική Βιομηχανία ένα στοιχείο το οποίο είναι ίσονο σημασία. Εξετάσαμε ε, τη δημιουργική βιομηχανία όχι μόνο για το πώς μας ενδιαφέρουν από οικονομική σκοπιά, αλλά για το τι επιρροή μπορούν να έχουν στην υπόλοιπη οικονομία είδαμε ότι η δημιουργική βιομηχανία έχει άμεση συνέπεια στους υπόλοιπους τομείς και στην ε, βιομηχανική οικονομία, γιατί αυτοί οι τομείς αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες από τον δημιουργικό τομέα και έτσι μπορούν να είναι πιο καινοτόμες. Και αυτό είναι ένα ε, μοναδικό στοιχείο. Ε, κάναμε και μία μελέτη βάσει της μελέτης αποδείχθηκε ότι σε κλίμακα βαλονίας ε, το 11% των προϊόντων ε, τα οποία παράγονται από τη δημιουργική βιομηχανία εντάσσονται ως ε, στοιχεία συνεισφοράς στους υπόλοιπους τομείς. Κυρίως ο αγροδιατροφικός τομέας, φαρμακευτικός και καλλιτικά προϊόντα. καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο δημιουργικός τομέας δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες που καταναλώνουν άλλοι τομείς. Το 11% δεν είναι πάρα πολύ μεν, αλλά είναι αρκετά ουσιαστικό δε. Υπάρχουν λοιπόν ε, αρκετά στατιστικά στοιχεία τα οποία μας καταδεικνύουν αυτά τα στοιχεία, αρκετά όρια, δεν θα σταθώ σε αυτά. Κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε ότι υπάρχει και ένα φαινόμενο ντόμινο. Ο δημιουργικός τομέας διαχέεται και στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργικός τομέας ε, παράγει γνώση και προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται από άλλες επιχειρήσεις, από άλλους τομείς και φαίνεται ότι υπάρχει μια επιστροφή προς αυτές τις δημιουργικές βιομηχανίες. Δεν θα πω άλλα γιατί θα καθυστερήσω και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η έμεση συνέπειες οι οποίες αφορούν ε, το δέλεαρ που μπορεί να έχει μια περιοχή όπως η Βαλονία και μπορούμε να τα δούμε και σε κλίμακα Μητρόπολης. Ε, μπορούμε να έχουμε σε κάποιους τομείς ε, και επιρροή σε άλλους οικονομικούς τομείς μιας περιοχής. Αυτά τα έχουμε και σε επίπεδο δικτύωσης, δημιουργούνται κλάστερς, ανταγωνιστικοί. Ε, τομείς που μπορούν να βοηθήσουν και να δημιουργήσουν ε, στοιχεία στη ε, δημιουργική βιομηχανία. Επίσης προσπαθούμε να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να συνεργαστούμε σε διάφορες διαστάσεις και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την συνεργασία μεταξύ της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και των υπόλοιπων τομέων και εδώ πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να εργαζόμαστε σε ένα οικοσύστημα γιατί δεν μπορούμε να δούμε τα στοιχεία μεμονωμένα και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα βλέπετε εδώ. Υπάρχει ένα μικρό βιβλίο το οποίο δυστυχώς ε, δεν διαθέτω σε πολλά αντίτυπα. Μπορώ να σας δώσω όμως ε, τον σύνδεσμο στο διαδίκτυο και μπορείτε να το λάβετε σε PDF. Ε, έχουμε τα αποτελέσματα που είχαμε, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2015 και είχαμε στοιχεία και για τη δημιουργική βιομηχανία, είχαμε συνεργασία μεταξύ δημιουργικής βιομηχανίας και άλλων επιχειρήσεων μέσω ενός συστήματος ε, τσεκ δημιουργικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα χρηματοδότησης για τη δημιουργική βιομηχανία και προσπαθήσαμε λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε και τον τραπεζικό τομέα για αυτή την πτυχή και θα έπρεπε να σταματήσω εδώ και ένα τελευταίο στοιχείο που αφορά αυτά τα clusters πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το δημιουργικό τομέα μέσω αυτών των κλάστερς με τον αγροδιατροφικό τομέα, με τον αεροναυπηγικό τομέα και πώς μπορούμε να έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το σχέδιο ή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να εργαστούν και σε άλλους τομείς. Δεν ξέρω αν ξεπέρασα το όριο των πέντε λεπτών. Έχω πολλές άλλες πληροφορίες για τη συνέχεια και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, καλά τα πήγατε. Έξι λεπτά και κάτι, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν εύκολο και σας ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να σας πω, δίνοντας το λόγο... για τους βουλευτές που δεν είναι στο πάνελ και θέλουν να ζητήσουν το λόγο, σας παρακαλώ συμπληρώστε το έντυπο που σας έχουμε δώσει και έτσι μπορούμε να σας συμπεριλάβουμε στον κατάλογο των αγορητών να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον και να δώσω το λόγο στον Πάτρικ Μπλος, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Γαλλίας, της, ε, της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι διότι σήμερα εκπροσωπώ την, Εθνική, ε, τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι τέτοιου είδους ανταλλαγές απόψεων μας εμπλουτίζουν και δίνουν νέα δυναμική στις διάφορες δράσεις. Αυτό είναι κάτι που έχω βιώσει ε, και διότι συμμετείχα στην... ήμουν παρόν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Μίδια του... Ε, της Γερμανικής ε, Βουλής. Σίγουρα η νομιμότητα των πολιτιστικών δράσεων ε, κατοχυρώνεται η νομιμοποίησή τους, κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες. Το καλλιτεχνικό και πολιτιστικό έργο δεν είναι εμπόρευμα. Έχει ιδιαίτερη φύση και άρα χρειάζεται να θεσπίσουμε ιδιαίτερο δίκαιο, ε, νομικές διατάξεις, προστατευτικές για να μπορούμε να έχουμε πάντοτε δημιουργία και ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Η Γαλλία ανέκαθεν Περασπιζόταν αυτή την αντίληψη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό είχε πει ανέκαθεν επιφυλεκτική στάση και ως προς το σχέδιο μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το, ε, στα θέματα των μίντια ή των ε, συγγραφικών δικαιωμάτων ε, πάντοτε είχαμε επιφυλακτική στάση και εναντί τη στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση τη TTIP. Στη Γαλλία, οι στρατηγικέ που έχουν κατα... αναπτυχθεί τα τελευταία ε, χρόνια είναι στρατηγικέ στήριξη των τομέων του πολιτισμού και τη δημιουργία και θεωρούμε ότι είναι στόχοι γενικού δημοσίου συμφέροντο. Και έχουμε τον νόμο τη 7 η Ιουλίου του 2016 για την ελευθερία τη δημιουργία την αρχιτεκτονική και την κληρονομιά. Και η λέξεις κλειδιά είναι ποικιλομορφία, ε, εγκύτητα, ανάπτυξη και ε, ε ανάμιξη. Ποικιλομορφία δημιουργών και έργων. Ο νόμος της 7ης Ιουλίου του 2016 επιβεβαιώνει στα δύο πρώτα άρθρα την ελευθερία της δημιουργίας και της καλλιτεχνικής διάδοσης των έργων. Αυτές οι διατάξεις μας επιτρέπουν να έχουμε ισχυρή νομική βάση για να αντιπαραταχθούμε στις τάσεις λογοκρισίας ή ελέγχου της πολιτιστικής ε, πρόσφορας. Ο νόμος ενισχύει τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και των συγγραφέων, των δημιουργών και συμπεριλαμβάνει εκεί και τους ψηφιακούς διάβλους διάδοσης του καλλιτεχνικού έργου. Το 2015 ε, στον νόμο έχουμε κατοχυρώσει τα δικαιώματα των ε, όσων έχουν προσωρινές συμβάσεις εργασίας και εργάζονται στο κινηματογράφο κυρίως και έχουμε ένα καθεστώς ασφάλισης και επιδομάτων ανεργίας που που προσαρμόζεται σε αυτού του είδους τα επαγγέλματα. Μιλούμε επίσης για την ανάμειξη του κοινού, δηλαδή να έχουμε κοινό από πολλές διαφορετικές ε, εθνοτικές ή άλλες καταγωγές. Η πρόσβαση στην τέχνη παραμένει άνηση, ισχυρά άνηση στην Ευρώπη και εμείς θέλουμε αυτό να το άρουμε. Θέλουμε ε, να ενισχύσουμε τη θέση και τα μέσα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής εκπαίδευσης και να ενισχύσουμε και την ερασιτεχνική τέχνη και την ερασιτεχνική, καλλιτεχνική και πολιτιστική δημιουργία. Μιλάμε επίσης για την εγκύτητα των χώρων πολιτισμού. Η πολιτιστική δράση των κοινοτήτων και των περιφερειών είναι απαραίτητη ε, την ε, πνευματική τροφή ε, τον ειδικότερα της υπαίθρου και έχουν γίνει σημαντικές ε, προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση κυρίως μέσω βιβλιοθηκών αλλά και βιβλιοθηκών οπτικοακουστικών μέσων. Μιλούμε επίσης για την ανάπτυξη της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας. Θέλουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που υφίστανται τον έντονο ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο και γι' αυτό ως Γαλλία έχουμε θεσπίσει ε, ενάρετους, ενάρετους μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης από τον ίδιο τον κλάδο για το κινηματογράφο και το οπτικοακουστικό τομέα, το ιδιωτικό θέατρο, το τραγούδι, το βαριετέ. Έχουμε ενισχύσει δηλαδή τους μηχανισμούς ε, απαλλαγών ή επιστροφών φόρου για να ενισχύσουμε τα γυρίσματα στη Γαλλία. Να γίνονται γυρίσματα στη Γαλλία ή να δημιουργούνται βιντεοπαιχνίδια στη Γαλλία ή να παράγονται μουσικά θεάματα που θα αναδεικνύουν νέα ταλέντα. Θέλουμε αυτό να έχει αποτέλεσμα στη δημιουργία πλούτου και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και πιστεύουμε ότι θα έχει όλα τα στοιχεία αυτό ε, δείχνουν. Θέλουμε να προωθήσουμε τον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό κλάδο, δηλαδή να διευκολύνουμε την κίνηση, να ενθαρρύνουμε τη δυναμική, το άνοιγμα, την περιέργεια και θα πρέπει οι καλλιτέχνε και τα έργα τους να είναι προσβάσιμα από παντού. Έτσι θα κινητοποιήσουμε, θα παρακινήσουμε και θα συγκινήσουμε ε, το κοινό όσο απομακρυσμένο και αν είναι από τον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σα και συγχαρητήρια και για αυτή τη νέα νομοθεσία που θεωρώ την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ε, Επίση, ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να μα δώσετε και το υλικό για να το διανύμουμε στου συναδέλφου. Τώρα να δώσω το λόγο στην Εντίτε Στρέλα, η οποία είναι εκεί κάτω. καλώ ορίσατε και παρακαλώ. Είναι πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού, Επικοινωνία, Νεολαίας και Αθλητισμού της ε, Πορτογαλική Δημοκρατία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, φίλη μου και πρώην συνάδελφό μου, θα ήθελα να πω ότι νιώθω συγκίνηση που βρίσκομαι πάλι εδώ στο Κοινοβούλιο, που πέρασα δέκα χρόνια της ζωής μου. Και χαίρομαι που μπορώ να επιστρέψω ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου της χώρας μου, της Πορτογαλίας. Η χώρα μου αποτελεί υπόδειγμα όσον αφορά τις επενδύσεις ε, στον πολιτισμό και τη δημιουργία. Ε, βασιζόμαστε στην ε, επιστήμη, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Αυτή η στρατηγική επιλογή έχει συμβάλει σημαντικά στις εξαγωγές της Πορτογαλίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα η πολιτιστική και δημιουργική τομή ε, είναι ε, ο τρίτος μεγαλύτερος τομέας ε, μετά τα τρόφιμα και τα ποτά όσον αφορά το, τη συμβολή τους στο ΑΕΠ. Θεωρούμε ότι τα αγαθά αυτά είναι πολύτιμα καταναλωτικά αγαθά. Οι καταναλωτές ψάχνουν κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Πριν λίγα χρόνια είχαν κατακλείσει την Ευρώπη προϊόντα χαμηλού κόστους από την Ασία και χρεοκόπησαν πολλές ε, επιχειρήσεις ρουχισμού ε, και υποδημάτων, διότι δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν το χαμηλό ε, κόστος της εργασίας στις χώρες της Ασίας. Γι' αυτό επικεντρώθηκαν σε προϊόντα υψηλής ποιότητας ε, και ε, καλέσει του σχεδιασμού. Δηλαδή σε προϊόντα ε, design και έτσι τα προϊόντα της Πορτογαλίας έχουν αρχίσει να αποκτούν μεγαλύτερο μερίδιο στις αγορές του κόσμου. Έχουμε τα δεύτερα πιο ακριβά παπούτσια στον κόσμο μετά τα Ιταλικά όσον αφορά τον εσωτερικό σχεδιασμό. Ε, έχουμε προβληθεί στο Hollywood και σε πολλές άλλες αγορές, σε πολλές πόλεις του κόσμου. Βλέπουμε έργα Πορτογάλων αρχιτεκτόνων. Δύο μάλιστα Πορτογάλοι αρχιτέκτονες ε, έχουν κερδίσει το βραβείο Πρίτσκερ που θεωρείται το Νόμπελ του, της αρχιτεκτονικής. Οι τομείς του πολιτισμού ε, αναπτύσσονται και δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Κάτι που επηρεάζει θετικά και τους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας μας. Πρόκειται λοιπόν ε, για μια νέα δομή. Ο πολιτισμός τροφοδοτεί την οικονομία. Ο πολιτισμός όμως είναι και μέρος ε, της ε, ταυτότητάς μας, της δημοκρατίας. Και πρόσφατα μόλις έχουν αρχίσει άνθρωποι και το συνειδητοποιούν αυτό και επικεντρώνονται στις κοινωνικές πτυχές του πολιτισμού. Για παράδειγμα υπάρχει το Μουσείο Guggenheim στο Bilbao που έχει βοηθήσει πολύ στην προβολή της πόλης αυτής σε όλο τον κόσμο και έχει βοηθήσει στην αναβάθμισή της. Ο πολιτισμός θεωρείται πια επένδυση και όχι απλά δαπάνη. Παρά τις ε, πιέσεις του προϋπολογισμού ε, έχουμε προσπαθήσει να επενδύσουμε στον πολιτισμό. Έχουμε δώσει δωρεάν πρόσβαση σε μουσεία κάποιες συγκεκριμένε μέρες. Είναι πολύ οικονομική είσοδος για τους ηλικιωμένους ή τους νέους. Υπάρχουν διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Πορτογαλία. Ε, επίση, έχουμε αλλάξει τι αρμοδιότητε του Υπουργείου Πολιτισμού και τα μέσα μαζική ενημέρωση τώρα πια υπάγονται σε αυτό. Και επίση ασχολείται το Υπουργείο Πολιτισμού και με το καθεστώ των ανθρώπων που εργάζονται ε, στα σχετικά επαγγέλματα. Επίσης ε, έχουμε διάδοση τη επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, περισσότερα κανάλια, τα οποία επιτρέπουν σε περισσότερο κόσμο στην Πορτογαλία να έρχεται σε επαφή με τον πολιτισμό. Επίσης δίδονται κάρτες πολιτισμού σε εργαζομένους, έτσι ε, έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά οι εργαζόμενοι και ε, η δαπάνη αυτή εκπίπτει από τη φορολογία για την επιχείρηση. Έχουμε προτείνει αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού για το 2017. Η αύξηση αυτή ε, συνάδει με το λογική της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και θα οδηγήσει σε ευφυή, βιώσιμη και συμμετοχική ανάπτυξη. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ενεργά να στηρίξει και να προωθήσει ε, τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς ε, στην Ευρώπη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά καθώς και τη γλωσσική μας κληρονομιά. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ανάγκες των τομέων αυτών και την ανάγκη να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην πρόσβαση για περισσότερο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το πλαίσιο το οποίο μας δώσατε, που είναι ε, και μία απόδειξη της πρόκλησης ε, της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης ε, που συνέβη και στη χώρα σας και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη νέα απασχόληση, την οικονομία και την καινοτομία. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Λουίτζι Μόργανο, επανειλημμένο σας ανέφερα ως εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να πω καταρχάς ότι δεν μπορώ να κάνω ε, κάτι για να σας ανακοινώσω το σχέδιο έκθεσης που εκπονούμε αυτή τη στιγμή. Επομένως θα σταθώ σε κάποια στοιχεία πολιτικής αξίας. Το πρώτο στοιχείο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ξεκινήσαμε από τα στοιχεία ε, για να προχωρήσουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης και να προτείνουμε και κάποιο πιθανό ορισμό με μία και μόνη έννοια. Την ε, λειτουργικότητα και την πρόσβαση στα κονδύλια χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα ερμηνείας τα οποία θα μπορούσαν ίσως ε, να ε, δημιουργήσουν και προβλήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ο πολιτικός στόχος αυτής της πρότασης, μια πρόταση που είναι κοινή της Ευρωπαϊκής ε, ε, της Επιτροπής Πολιτισμού και της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Έξι χρόνια μετά το ε, πράσινο βίβλο πρέπει να δοθεί ένα άλμα ποιότητας και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής συνεκτικό και μακροπρόθεσμο για τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία που να προωθεί την ε, τις βιομηχανίες αυτές και να τις προστατεύει και να θεωρείται στρατηγικός στόχος και πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά γιατί ο πολιτισμός, η τέχνη, η δημιουργικότητα και η ομορφιά είναι πρώτη ύλη της Ευρώπης και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην ε, ψηφιακή μετάβαση η δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία σταδιακά αντικαθιστούν ε, τις γραμμές παραγωγής και τις ε, ε, αλυσίδες αξίας που είχαμε στο παρελθόν, όπως πολύ σωστά επεσήμαναν όσοι μίλησαν πριν από μένα. Δεύτερον, η διτή αξία, η οποία συνδέεται άρρηκτα με αυτές τις πραγματικότητες. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες είναι ένα εργαλείο για να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε την γλωσσική και πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης, να ενισχύσουμε την ποικιλομορφία ομορφία της Ευρώπης και να προωθήσουμε την άειλη και ηλική πολιτιστική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενοές. Ταυτόχρονα όμως είναι και πάρα πολύ σημαντικές για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, λαμβάνοντας υπόψη και την ε, μεγάλη συνεισφορά που έχουν στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλό δε μάλλον γιατί υπάρχουν και συνέπειε καινοτομία σε άλλου τομείς όπω τον τουρισμό, το λιανεμπόριο αλλά και την ε, ψηφιακέ ε, οικονομίες. Ε, επίσης, ε, αυτά διαδραματίζουν πολύ σημαντικό στην ευρωπαϊκή πολιτιστική ε, βιομηχανία για να ενισχύσουμε τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Να αποτελούν δηλαδή την ήπια δύναμη της Ευρώπης ώστε η δημιουργικότητα, η αριστεία, η βιοτεχνία, ο πολιτισμός, όλα αυτά μας θέτουν στο προσκήνιο παγκοσμίω. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη ε, από πλευράς πολιτικής και να δοθεί μια συγκεκριμένη απάντηση, διότι θα αποτελέσει απάντηση και στην κρίση, κυρίως ε, στην κρίση ενεργείας των νέων. Εάν όπως υποστηρίζει η πλειοψηφία των συναδέλφων αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό το θέμα της ανεργίας των νέων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να επιλύσουμε και είναι από τους βασικούς στόχους της Ευρώπης, κάθε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει ως στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας ποιότητας και επομένως υπάρχει ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό εδώ. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι απασχολούν πάνω από 12 εκατομμύρια εργαζομένους με πλήρη απασχόληση, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωση και δημιουργούν ένα κύκλο προστιθέμενης αξίας 500 δι ευρώ στην ε, στο ΕΕ της Ένωσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κατά πόσο θα πρέπει να διευρυνθεί ή όχι είναι άλλη συζήτηση, αλλά θεωρώ ότι το στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, η ίδια η επαναβιομηχώνηση της Ευρώπης, που είναι ένα στοιχείο το οποίο ιδια η επαναδιαμηχωνηση της ευρωπης που ειναι ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και εμάς, σίγουρα περνάει από πολιτικές οι οποίες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις μεγάλες δυνατότητες αυτών των κλάδων. Και γιατί αυτό. Διότι σαφέστατα υπάρχουν μια σειρά από θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στον τομέα της ανάπτυξης, στον τομέα της σχέσης μεταξύ επένδυσης και επιστροφής ε, της επένδυσης και φυσικά και για άλλους ε, βιομηχανικούς τομείς όπως ε, ο τουρισμός, οι ψηφιακές τεχνολογίες και το λιανικό εμπόριο. Ένα ε, περαιτέρω ζήτημα εδώ, το οποίο έχει σχέση και με τους άλλους κλάδους, είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Στις συγκεκριμένες βιομηχανίες εργάζονται περισσότεροι νέοι, μεταξύ 19 και 29 ετών, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο οικονομικό κλάδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι, για παράδειγμα, είναι 2,5 φορές περισσότεροι από την αυτοκινητοβιομηχανία και 5 φορές περισσότεροι από τη χημική βιομηχανία. Κατά μέσο όρο είναι κατά 2 φορές ανώτερο από όλο τον τραπεζικό τομέα και τον ασφαλιστικό τομέα. Η πλειοψηφία των κλάδων αυτών αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, λιγότερο από 9 υπαλλήλων δηλαδή. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ελήφθη υπόψη και είναι πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού, διότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του όλου κλάδου αυτή τη στιγμή και επίσης η συγκεκριμένη κλάδη δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο 90% του εργατικού δυναμικού τους είναι ε, ε, επιχειρήσεις που έχουν κάτω από 9 υπαλλήλους. Και ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό ήταν αυτές οι οποίες προσαρμόστηκαν πολύ καλύτερα στην οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε το 2008. Εδώ σας λέω επιγραμματικά μόνο τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναπτύξω στην έκθεσή μου διότι έχω καθυστερήσει. Υπάρχει το θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης το οποίο πολύ σωστά επισημάνατε. Επίσης υπάρχει και ορισμός ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως πρόταση ε, αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει συγκεκριμένε παραμέτρου, οι οποίε πρέπει ε, να βοηθούν να ερμηνεύονται επακριβώ τα στοιχεία. Δεν υπάρχει λόγος ε, να ε, τιμωρούνται άλλοι παραδοσιακοί τομείς λόγω τη ασάφεια ενό ορισμού. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να υπάρξουν και παρανοήσει οι οποίε δεν θα έπρεπε να έχουν. Οι παραδοσιακοί τομεί, όπω μουσεία, βιβλιοθήκε, φεστιβάλ κλπ. θα πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη οικονομική χρηματοδότηση με κονδύλια τα οποία θέλουν να βοηθήσουν τη συνέχεια και την ανάπτυξή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λάβουν υπόψη και την άλλη πτυχή, διότι η ενίσχυση των πολιτικών και νομοθεσία που σχετίζεται με την πνευματική ιδιοκτησία, την καταπολέμηση ε, των... Ε, παραποιημένων αγαθών και επίσης το να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και νέα ταλέντα ε, είναι ε, πολύ σημαντικά στον τομέα της μόδας και της βιομηχανίας υψηλής πότητας. Τα υπόλοιπα την άλλη φορά. Ε, βλέπετε το θέμα είναι ευρύτατο διακόπτη πρόεδρο στον ομιλητή και είναι πολύ δύσκολο να συνοψίσουμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο πρώτα στους προσκεκλημένους μας, στους εθνικούς βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο και μετά στους ευρωβουλευτές ε, Ιζαμπέλα Χέκμαρκ από τη Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος. Ε, δύο λεπτά ο καθένας σας παρακαλώ, όχι περισσότερο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ε, παρουσιάσεις που ακούσαμε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να πω για τους δημιουργικού ε, τομείς ότι θα πρέπει να βασίζονται στην καινοτομία, αλλά όχι στα παλιά μοτίβα τα οποία ούτως ή άλλως στηρίζουν οι πολιτικοί. αν πιστεύει κανείς ε, ότι θα μπορούσε ε, η πολιτική να χρηματοδοτήσει το Spotify, ε, για παράδειγμα, μάλλον κάνει λάθος. Άλλο παράδειγμα είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που πριν μερικά χρόνια θεωρείται ότι αντίκυνταν στα, στους πολιτιστικούς εθνικούς στόχους οι περισσότερες ε, μορφές ε, ενίσχυσης ε, στηρίζουν τα παλιά μέσα που γνωρίζουμε και με παλιές κλίδες κατανομής. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Πώς μπορούμε να φροντίσουμε να έχουμε νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων που να στηρίζει τους νέους, τους μικρούς και τις ψηφιακές επιχειρήσεις για να δημιουργηθούν και νέες μορφές κατανομής. Ευχαριστώ. Μπέλα ντομάντα. Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, γι' αυτό να πω ότι ανάλογα με την παρέμβαση θα απαντήσει και κάποιος, αλλιώς θα προσπαθήσουμε και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υποφαινόμενη να σας απαντήσουμε. Η κυρία Λεούτσι από την Ιταλία, από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ο κύριος Λεούτζη, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα, διότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση και φυσικά έχουμε αυθεντίες που το συζητούν. Δύο-τρεις σκέψεις. Τα μουσεία πρέπει να πάψουν να είναι μουσεία και οι πινακοθήκες πρέπει να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Πρέπει οι χώροι αυτοί να πάψουν να είναι χώροι της ελίτ που απευθύνονται μόνο στους λίγους ε, πρέπει και μέσω της δημιουργικής βιομηχανίας να δοθεί περισσότερος χώρος στην τεχνολογική καινοτομία και να προσεγγίσουν τους λαούς και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και ε, φυσικά των υπηρετικών κοινοτήτων. Να πω και δύο λόγια για τα λεγόμενους ε, τρόπους εγκατάληψης. Αναφέρθηκε εδώ και η ε, βιομηχανική αρχαιολογία. Ε, υπάρχουν κατάλληλε πηγές ενδιαφέροντος και συνεπώς και απασχόλησης ε, στα πλαίσια μιας απόπειρα ε, να αναδιοργανώσουμε και να ανανεώσουμε όλους αυτούς τους χώρους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται πλέον και θα μπορούσαν να γίνουν χώροι της δημιουργικότητας και να μας επιτρέψουν να έχουμε νέες εξελίξεις και νέες ευκαιρίες και για την ε, απασχόληση των νέων. Αυτό είναι έκκληση βέβαια που σας κάνω. Αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από κάποιες εβδομάδες στην Ιταλική Γερουσία, που ομόφωνα, σχεδόν ομόφωνα, εγκρίθηκε μια ε, πρόταση την οποία δέχθηκε η κυβέρνηση για να παρέμβει για να ε, χρησιμοποιηθούν οι λεγόμενοι τίτλοι τέλους ε, των τηλεοπτικών εκπομπών σε ιδιωτικές και τηλεοπτικές τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Στους τίτλους τέλους αναφέρονται τα διάφορα επαγγέλματα, ε, τα δημιουργικά επαγγέλματα, βιοτέχνες, άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν και συμμετέχουν ε, στη δημιουργία ενός ε, κινηματογραφικού έργου. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή ξεχνιούνται για να υπάρχει χώρος για τη διαφήμιση, ενώ κανονικά θα πρέπει να προβάλλονται καταλήλως για να μπορούν και αυτά τα επαγγέλματα να προβάλλονται όσο πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε έναν Έλληνα βουλευτή τώρα από την ΚΟΕ. Νικόλος Θηβαίος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος. Η Ελλάδα παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει σε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική δραστηριότητα με οδηγό μια πλουραλιστική, πολυπολιτισμική και κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική. Στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής δραστηριοποιούνται άμεσα ή επικουρικά θεσμοί πολιτισμού, εκπαίδευσης, τουρισμού από την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, ομάδες πολιτών δημιουργών, δομές αλληλεγγύης με φροντίδα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα με αφορμή τη συνάντησή μας θα ήθελα να αναπτύξω ιδιαίτερα το θέμα νέοι δημιουργοί στην Ελλάδα. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι στη χώρα μας δημιουργούν και επιχειρούν μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες με κύριο πρόβλημα την ανέβρεση κτηριακών υποδομών και μέσων ικανών να στεγάσουν, να προβάλλουν και να αναπτύξουν τη δημιουργική τους προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα νέοι ηθοποιοί, μέλη θεατρικών ομάδων, καθώς και μουσικοί, προσπαθούν να στεγάσουν τη δημιουργική τους προσπάθεια. Για τη στέγαση τέτοιων δημιουργικών σχημάτων στην Ελλάδα μπορούν να αξιοποιηθούν ιστορικά κτίρια, κτίρια με ιδιαίτερη κοινωνική αξία, αποθήκες, παλιοί κινηματογράφοι. Η αξιοποίηση πολλές φορές με λίγα χρήματα τέτοιων χώρων θα έδινε τεράστια όθηση στην πολιτιστική δημιουργία, στην επαγγελματοποίηση του τομέα και την βελτίωση της ποιότητα των έργων των νέων δημιουργών. Επίση, θα ήταν χρήσιμο και για του νέου δημιουργούς αλλά και γενικότερα για τον πολιτιστικό αγαθό, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει μια στρατηγική επικοινωνία και ανταλλαγή πολιτιστικών δράσεων, ένα πολυδιάστατο δηλαδή πολιτιστικό εράσμου που θα δώσει νέε δυνατότητε, ευκαιρίε και ιδέε για πολιτισμό και δημιουργία. Σε αυτόν τον τομέα βέβαια σημαντικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν τόσο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα εθνικά κοινοβούλια σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι αναγκαία η αύξηση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθεται και τον πολιτισμό και τον δημιουργικό τομέα μέσω ευέλικτων προγραμμάτων στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ζητηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του νέου εγχειρήματο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για αυτή την τελική σας έκκληση που νομίζω ότι βρίσκει πολλούς σύμφωνους. Μπαρτ Κάρον τώρα από το Βέλγιο, από τους Πρασίνους, παρακαλώ. Συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ. Είμαι βουλευτής ε, του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου και πιστεύω και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα οι επενδύσεις ε, στην πολιτιστική καινοτομία και πολυμορφία. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά βασίζονται και στην τέχνη και σε τομέα που δεν αποφέρει κέρδος. Τα δύο αυτά μαζί όμως επιφέρουν προσθέμενη αξία ε, στην οικονομία και την κοινωνία. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μία έκκληση. Την ε, τέχνη και τον πολιτισμό, να μην τα θεωρήσουμε μόνο υποτομέα της οικονομίας, ε, αλλά να τα θεωρήσουμε και ανεξάρτητο τομέα. Η Φλάνδρα και οι κάτω χώρε ε, είναι η επίσημη προσκεκλημένη χώρα, η τιμόμενη χώρα στην ε, έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης. Οι συγγραφείς και οι μεταφραστές μας εποφελούνται από κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό για την οικονομία. Η κυβέρνηση της Φλάνδρας ε, στηρίζει τις δράσεις αυτές. Τέλος θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για την δημιουργική οικονομία αλλά και για την τέχνη και για τους καλλιτέχνες. Δεν θα πρέπει ο πολιτισμός ε, να ε, ακολουθεί την οικονομία ή το αντίθετο. Θα πρέπει μαζί να στηρίξουμε και τα δύο. Ευχαριστώ. Να πω απλώς ότι εμείς συμφωνούμε απολύτως ο τίτλος μάλιστα είναι «Δημιουργική και πολιτιστική κλάδη». Ε, η πολιτιστική βιομηχανία είναι μία πτυχή, αλλά ε, αναφερόμαστε σε θέματα τα οποία έχουν αυτή τη διπλή φύση, πολιτιστική και οικονομική, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη διευκρίνηση. Να δώσω τώρα το λόγο σε τρεις συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να σας πω απλώς ε, ότι θα μπορούσατε να παρέμβατε και στα άλλα πάνελ, γιατί φαίνεται να συγκεντρώνεστε εδώ και να καθυστερήσουμε λίγο στο πρώτο πάνελ μετά στη συνέχεια. Η Πέτρα Κάμερ Εύερτ, συντονίστρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Επιτροπή Πολιτισμού. Παρακαλώ, Πέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις που ακούσαμε μέχρι τώρα. Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση προς τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όλα γνωρίζουμε το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe. Ξέρουμε όμως και τις περιορισμένες δυνατότητες του προγράμματος αυτού, διότι δεν χρηματοδοτείται με αρκετά χρήματα για να αποτελέσει επαργή προώθηση ε, του πολιτιστικού τομέα. Αλλά λόγω και της πίεσης ε, της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στην ε, για τη νέα περίοδο ε, έχουμε δημιουργήσει δυνατότητες ε, μέσω των διαφθορτικών ταμείων, ώστε να διατίθενται πόροι για προώθηση ε, του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Και θα με ενδιέφερε σε τι βαθμό στα κράτη-μέλη δαπανώνται τα χρήματα, διότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για τα διαρθρωτικά ταμεία. Δηλαδή χρησιμοποιείται περισσότερο αυτή η δυνατότητα διότι μπορεί να αποτελέσει έναν καλό τρόπο από τη μία μεριά να καταπολεμήσουμε την ε, ανεργία αλλά να προωθήσουμε και τις ε, πολιτιστικές και δημιουργικές ε, δράσεις ταυτόχρονα. Θα με, διέφερνε, θα με λοιπόν να μάθω εάν αυτή η δυνατότητα που δημιουργήσαμε πράγματι χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη. Ίσως και η Κομισιόν να έχει σχετικές γνώσεις. Ωραία. Υπάρχει αυτή η ερώτηση. Όποιο θέλει την απαντά στη συνέχεια, όσο θα τη σκέφτεστε, να δώσω το λόγο στην κυρία Χέλγα Τρούπελ, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού από τους Πρασίνους. Παρακαλώ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, σας θυμίσω την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης ε, του Προέδρου Γιούνκερ που αναφέρθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία θέλει να δημιουργήσει μια ψηφιακή εσωτερική αγορά, από την άλλη χρειάζεται ε, επιγόντως ε, δίκαιη αμοιβή των καλλιτεχνών στο επιγραμμικό περιβάλλον. Και θίξατε εσείς το ερώτημα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω ότι επιγόντως χρειαζόμαστε ορισμό ώστε οι επιγραμμικές πλατφόρμες ε, να καθορίζουν το περιεχόμενο και να μην ε, είναι απλά ε, οι υπηρεσίες μετάδοσης, διότι αν είναι αυτό τότε δεν φέρουν ευθύνη. Είναι σαφές όμως ότι δεν είναι τόσο ουδέτερες αυτές οι υπηρεσίες, αλλά οργανώνουν το περιεχόμενο. Η διάκριση όμως ανάμεσα σε έναν ουδέτερο φορέα και έναν που οργανώνει το περιεχόμενο, χρειαζόμαστε σωστό ορισμό. Θα ήθελα λοιπόν από την Κομισιόν αλλά και από εσά, ε, συναδέλφοι από τεχνικά κοινοβούλια, να μάθω εάν κάποιο εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό ή αν υπάρχουν ιδέε για το πώ μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και χαίρομαι που το έφυξες η Julie Ward και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ, εκτός και αν υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις από αυτή την πλευρά. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να απαντήσω στον βουλευτή που ρώτησε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις ή τους μεμονωμένους καλλιτέχνες που μόλις ξεκινούν ε, τη σταδιοδρομία τους. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά η δικτύωση και οι οργανώσεις είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος να γίνει κάτι τέτοιο. Στην ε, δική μου περιφέρεια, στα βορειοδυτικά της ε, Αγγλίας, έχουμε μια εξαιρετική τέτοια οργάνωση, όπου νέοι αναδυόμενοι καλλιτέχνες συναντώνται. σε εργαστήρια, σεμινάρια σε μια κοινή προσπάθεια, ώστε να μην χρειάζεται οι καλλιτέχνε να περνούν το χρόνο του συμπληρώνοντα γραφειοκρατικά έντυπα. Και είναι ένα τρόπο να ενδυναμώσει κανεί του ανθρώπου αυτού, να του δώσει αυτοπεποίθηση, να του δώσει μια φωνή. και τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν ε, τα προβλήματα που, ε, ε, με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ένας νέος καλλιτέχνης. Οι καλλιτέχνε και αυτές οι οργανώσεις ε, πολύ συχνά λειτουργούν καλά όταν ε, υιοθετούν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως είναι οι συνεταιρισμοί. Και όσον αφορά το θέμα των άδειων κτηρίων, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα που αναγνωρίζουν ότι οι καλλιτέχνες συχνά έχουν μεγάλο πάθος για τη δημιουργία και μικρές χειρονομίες μπορούν να τους βοηθήσουν πάρα πολύ. Αν βρούμε τρόπου, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε υπάρχοντες ε, πόρους, διότι οι καλλιτέχνες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά με πολύ ενδιαφέροντε τρόπους. Είδαμε λοιπόν ε, εξαιρετική χρήση παλιών βιομηχανών κτηρίων σε πολλέ από τι πόλεις μα. Θα ήθελα πολύ να δω αξιοπρεπεί πολιτικέ για κάτι τέτοιο, ώστε ε, τα κενά κτίρια και οι καλλιτέχνε που τα χρησιμοποιούν να αποτελέσουν μέρο τη κυκλική οικονομία, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο παρουσιάσεων. Θα ήθελα να σας ζητήσω να δώσουμε προτεραιότητα στον συντονιστή της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης ε, πριν από τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατί πρέπει να φύγει, τον κύριο Μπόγκταν Βέντα από το ΕΛΚ, εισηγητής ε, του, ε, μιας εξαιρετικής έκθεσης, ο Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή και παρακολουθεί τις εργασίες φυσικά της Επιτροπής μας. Στη συνέχεια έχουμε τη Χάιτι Πούργα από την Εστονία, το Φλωρίνα Αλεξάνδρου Αλέξε από τη Ρουμανία, και την κυρία Χέρλιν Γκούντελαχ από τη Γερμανία. Παρακαλώ, Μπόκταν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ως μέλος της Επιτροπής Ήμουνα εισηγητής ε, της έκθεσης ε, για τις ευρωπαϊκές ταινίε στην, στην ψηφιακή εποχή. Ε, κάποια από τα σχόλια αφορούν και αυτό το τομέα και θα, έπρεπε να τα, θα ήθελα να τα λάβω υπόψη και πραγματικά εκτιμώ την παρέμβασή σα. Τώρα είμαι σκιώδη εισηγητή για τη δημιουργική βιομηχανία εκ μέρου του ΕΛΚ και θεωρώ ότι δεν αναγνωρίστηκε η σημασία του ε, δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα δεόντως από την πολιτική. Οι, τομεί αυτοί, οι τομείς αυτοί καθοδηγούνται από τον ίδιο στοιχείο, από τη δημιουργικότητα. Ε, είναι μια ελεύθερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που αυθονεί στις χώρες μας. Η δημιουργικότητα τροφοδοτείται από τον πολιτισμό με την ευρεία έννοια. Αυτά τα στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι ένα κοινό αγαθό τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε. Στη δεκαετία του 90 η Ευρωπαϊκή Ένωση βίωσε μια τεράστια αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων ε, της δημιουργικής βιομηχανίας και έτσι δημιουργήθηκαν και πολλές θέσεις εργασίας. Και αυτό φυσικά έχει σχέση και με την ποικιλομορφία μας. Ε, η δημιουργική βιομηχανία βοηθά στην ανάπτυξη των ε, τεχνολογιών πληροφορικής που είναι πάρα πολύ σημαντικές τεχνολογίες και για τις περιφέρειες και για τις χώρες και για το σύνολο της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τη δημιουργικότητα των ε, ε, δημιουργών μας ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τις δημιουργικές επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια εταιρική σχέση και αυτό σημαίνει ε, μόνιμη διαβούλευση με τους εκπροσώπους του κλάδου. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη του τομέα αυτού και να ε, μην υπάρχουν προσκόμματα στην ε, κινητικότητα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη των δημιουργικών βιομηχανιών σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να υπάρχει στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς και ε, ε, σε συγκεκριμένες αλλαγές ε, στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, κατάλληλη φορολόγηση ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να πάρουμε χρηματοδότηση από διάφορα ταμεία ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν καταλήτη ώστε να υπάρχουν και δυνατότητες ε, και κατάλληλη προσαρμογή του φορολογικού συστήματος θα μας το επιτρέψει αυτό. Ο κύριος Μόργανο αναφέρθηκε και σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και προσδίδει ελπίδα, αλλά παρεμβαίνει και ε, στο πολιτιστικό προσκήνιο. Υπάρχουν διάφορες μορφές διανομής και τα θέματα πνευματικού, πνευματικών δικαιωμάτων ε, είναι κάτι το οποίο δεν απασχολούν αυτή τη στιγμή τους καταναλωτές. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες των τομέων αυτών πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη εκπαίδευση ποιότητας σε πολύ ψηλό επίπεδο του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στις τεχνολογίες, πρέπει να υπάρχει προστασία από τις μεγάλες ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες πολλούν πολιτισμό σε τιμές ευκαιρίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πει και πολλά δυστυχώς στον τομέα αυτό, αλλά ε, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των προκλήσεων με τη συνεργασία των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Μπόγκταν. Ξέρουμε ότι πρέπει να φύγεις. Ε, εάν μπορέσει να παραμείνεις θα χαρούμε βεβαίως. Να δώσω τώρα μέσω στο λόγο στην κυρία Χάιντι Πούργα, μέλον της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Παιδείας από την Εσθονική Βουλή. Παρακαλώ. <laughs> Please Εκτός μικροφώνου. Good afternoon. Καλησπέρα σας. Είμαι μέλος της ε, Επιτροπής Πολιτισμού της Εσθονικής Βουλής. Ανήκω στο κόμμα των μεταρρυθμιστών που ανήκει στην πολιτική ομάδα του Άλτε, των Φιλελεύθερων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας μιλήσω για το πώς έχει η κατάσταση με τη δημιουργική βιομηχανία στην Εστονία, η οποία αναπτύσσει αυτό το κλάδο της οικονομίας συνειδητά από το 2004. Κάναμε χαρτογράφηση του κλάδου και είδαμε πόσοι απασχολούνται ε, και πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν. Έχει αυξηθεί ο αριθμός τους με την πάροδο των ετών και οι επιχειρήσεις έχουν γίνει όλο και πιο μικρές. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να έχουμε στρατηγική χρήση και στρατηγικό σχεδιασμό όλων των βιομηχανιών. Σήμερα τα ποιοτικά προϊόντα και η πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα και σε υποδομές είναι ο κανόνας στην Ευρώπη. Ε, οι άνθρωποι επιλέγουν συγκεκριμένο προϊόν, συγκεκριμένο χώρο να κατοικήσουν, ε, συγκεκριμένο κλάδο να δραστηριοποιηθούν για προσωπικούς λόγους, ο σύγχρονος καταναλωτής είναι πολύ πιο έξυπνος, πιο συνειδητοποιημένος ε, από οτιδήποτε πριν. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι πώς η Εστονία μπορεί να διατηρήσει τη, τη βιομηχανία της δημιουργίας στο επίκεντρο. Έχουμε αύξηση της ενσυναίσθησης, της συνειδητοποίησης, προσφέρουμε κατάρτιση, στηρίζουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις εξαγωγές. Θέλουμε να αναπτυχθεί η δημιουργική βιομηχανία με το πνεύμα της επιχειρηματικότητας. Είναι πολύ σημαντική η κλάδη αυτή γιατί κάνουν τη χώρα μας πολύ πιο ανταγωνιστική διεθνώς. Ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα διανοητικής ε, ιδιοκτησία, την καινοτομία, τα διπλώματα ευρεσιταχνία, είναι ε, δράσεις που θέλουμε να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε. Έχουμε παραδείγματα με επιχειρήσεις που ασχολούνται με την καθαρή γεωργία, με τη δημιουργία ε, δημιουργικών καινοτόμων προϊόντων με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ωφελούν τη χώρα γενικότερα, ούτως ή άλλως, και πιο συγκεκριμένα περιοχές της Εσθονίας. Προωθούμε την τοπική κουλτούρα ε, αυτό έχει σημασία σε περιφερειακό επίπεδο γιατί οι σφίζουσες από ζωή περιφέρειες προσελκύουν τους ανθρώπους και αξιοποιούμε την πολιτιστική κληρονομιά για την ανάπτυξη κάθε περιφέρειας. Έχουμε ε, φεστιβάλ ε, κινηματογράφου, φεστιβάλ μουσικής, όλα αυτά έχουν γίνει πραγματικά συνήθειες δεκαετιών έτσι εμπλέκονται όλο και περισσότεροι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και ελαφρύνεται το κράτος, δεν χρειάζεται να επενδύσει τόσο πολύ. Είναι εκδηλώσεις και γεγονότα που διαμορφώνουν τον ε, τομέα τον ακουστικό και τον κλάδο της μουσικής στην Εστονία εν γέννη. Να σας πω δύο λόγια και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ο τομέας της τεχνολογίας έχει πραγματικά ιστορίες επιτυχημένες να επιδείξει, success story, αλλά αυτό δεν αρκεί για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Δεν ακολουθούμε τη λογική των νεοφιών επιχειρήσεων στην τεχνολογία. Έχουμε σταθερές επενδύσεις σε βάθος χρόνου για να έχουμε ταλέντα, να αναδείξουμε ταλέντα από την αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας ή από την αρχή των σπουδών τους. Οι στόχοι μας είναι διτί, Πρώτον, οι επιχειρήσεις ε, που ανήκουν στην δημιουργική βιομηχανία να μπορούν να επιτύχουν σε συνθήκες αγοράς. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος και γι' αυτό αξιοποιούμε τα σχετικά εργαλεία. Και δεύτερον, η δημιουργική σκέψη θέλουμε να καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχουν οι Εστονοί και οι εστονικές επιχειρήσεις. Έτσι δημιουργείται προστιθέμενη αξία για κάθε απασχολούμενο. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και η γενική και η ειδική εκπαίδευση ε, είναι ευκαιρία για να ενισχύσουμε την εγχώρια κατανάλωση προϊόντων πολιτισμού. Και πρέπει ως προς την ανώτατη εκπαίδευση να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο οι διάφοροι κλάδοι να λεπιδρούν μεταξύ τους. Το σχέδιο, ο κλάδος του design με τις υπηρεσίες υγείας, με τη μηχανολογία και το καθεξής. Δηλαδή, είναι κλάδοι της οικονομίας πολυεπίπεδη, πολυδιάστατη και μπορούν να συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι άνθρωποι δεν επιλέγουν πλέον ένα προϊόν, αλλά προτιμούν μάρκες που έχουν μια ιστορία να πούν, που φέρνουν μαζί τους συναισθήματα επίσης και ιδέες και έννοιες. Η κατανάλωση δεν έχει να κάνει με την κάλυψη των βασικών αναγκών μας πλέον, αλλά είναι μια δήλωση κουλτούρας, αυτό που επιλέγει ο καθένας να καταναλώσει το κράτος έχει αρχίσει να πιστεύει σε αυτούς τους κλάδους και να επενδύει σε αυτούς. Σίγουρα η οικονομική κρίση είχε αντίκτυπο σε αυτό το κλάδο της οικονομίας, ωστόσο μπορούμε να αναπτυχθούμε περισσότερο. Μπορούμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, να έχουμε χορηγίες, να προωθήσουμε το μάρκετινγκ, να έχουμε ομάδες στόχους τις οποίες θα ε, ενισχύσουμε. Όλα αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Φλόριν Αλεξάνδρου Αλέξη από τη Ρουμανία, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και των Μέσων Ενημέρωσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τη θεσμική συνένεση όσο ό,τι αφορά τα, επιχειρη... επιτυχημένα επιχειρηματικά project. Πρόκειται για το φεστιβάλ Ιονέσκου που είναι ένας μεγάλος συνθέτης που αποβίωσε το 1955. Έζησε στη Γαλλία, στην Αυστρία και στη Ρουμανία. Ήξερε πολύ καλά τη μουσική γλώσσα ε, του 20ου ε, αιώνα. Μεγάλος συνθέτης, μεγάλος ε, βιολονίστας και πιανίστας. έλεγε ότι ως δάσκαλος αυτή ήταν η παράμετρος βάση της οποίας έκρινε όλους τους άλλους. Ε, και κυρίως η ιδιότητα του μαθητή ήταν αυτή που τον επηρέασε σε όλη του τη ζωή. Έχουμε λοιπόν το φεστιβάλ Ιονέσκο ε, από το 1958, κάθε τρία χρόνια ε, στην αρχή, κάθε δύο χρόνια μετά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μουσικά φεστιβάλ. Το 2015 το φεστιβάλ διάρκησε 22 ημέρες και δόθηκαν περίπου 58 συνευλίες ενώ πουλήθηκαν πάνω από 50.000 εισιτήρια, αλλά και άλλες πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις διοργανώθηκαν παράλληλα, όπως το Creative Bucharest, το Δημιουργικό Βουκουρέστι, και είχαμε πολύ σημαντικούς διεθνείς δημιουργούς που προσκλήθηκαν και έδωσαν το παρόν, αλλά και διάσημους μαέστρους και διάσημες ορχήστρες, η φιλαρμονική του, Βερολίνου, η ορχήστρα του Άμστερνταμ, η φιλερμονική του Ισραήλ, η συμφωνική ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο μεταξύ άλλων. Τέτοιου είδου εκδηλώσει δεν μπορούν να γίνουν χωρί θεσμική και οικονομική στήριξη. Εξού και ψηφίστηκε σχετικό νόμο το 2002 που ε, καθορίζει τη διοργάνωση και του τρόπου χρηματοδότηση αυτού του φεστιβάλ. Ο ίδιο ο πρόεδρο ε, θέτει ε, το φεστιβάλ υπό την αιγίδα του και το φεστιβάλ χρηματοδοτείται κυρίω από το Υπουργείο Πολιτισμού τη Ρουμανία. Την διοργάνωση του φεστιβάλ αναλαμβάνουν στελέχη των διαφόρων υπουργείων. Παρόλα αυτά κατά από τη στιγμή που το φεστιβάλ έγινε πολύ μεγάλο, συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η διοικητική δομή και διοργανωτική είναι κάπως δίσκαμπτη και γι' αυτό η Εθνική Τηλεόραση και το Εθνικό Ρουμανικό Πολιτιστικό ε, Ινστιτούτο έχουν αναλάβει τη διοργάνωσή του μαζί με δύο επαγγελματίες, εταιρείες δηλαδή επαγγελματικές εξειδικευμένες στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αλλά και το, το, οι δημοτικές αρχές του Βουκουρεστίου είναι ε, μέλος πλέον στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο, να το πω έτσι, που διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ. Η κυβέρνηση εγγυάται τη χρηματοδότηση. Ενώ το R-Cube που είναι η μία ε, ε, εταιρεία διοργάνωσης ασχολείται με την εξέβρεση των καλλιτεχνών και η άλλη εταιρεία διοργάνωσης ασχολείται με τη σύναψη των συμβάσεων. Είναι ένα φεστιβάλ εξαιρετικά σημαντικό για την εικόνα του Βουκουρεστίου και της χώρας μας εν γέννη. Το Βουκουρέστι έχει ωφεληθεί τα μάλα από τη διοργάνωση αυτής της καλλιτεχνικής εκδήλωσης. Ε, παράλληλα και άλλες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν παράλληλα με το φεστιβάλ Ενέσκο και νομίζουμε ότι είναι υπόδειγμα, είναι πρότυπο ε, που μπορεί να ακολουθηθεί και από άλλους για τη σύναψη συμμαχιών ε, στα μεγάλα καλλιτεχνικά project, γιατί έχει θεαματικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο να ακούμε να μιλάει κάποιος για μουσική και τώρα ο κύριος Γκούντελαχ, από πρόεδρος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης από τη Γερμανία. Πέντε λεπτά και πάλι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Η οικονομία του πολιτισμού και της δημιουργίας ε, στην ε, Γερμανία θεωρείται κεντρικός οικονομικός τομέας για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Παρ' όλα αυτά, ε, περνάει μεταβολή ο τομέας αυτός και η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει αφήσει εμφανή σημάδια και οι ε, συνθήκες πλαίσιο ε, έχουν αλλάξει λόγω της διεθνοποίησης. Η μεταβολή αυτή έχει οδηγήσει στο να εμφανιστούν νέοι παράγοντες και να έχουμε πολύ μεγάλες και πολύ μικρές επιχειρήσεις δίπλα-δίπλα. Οι αλλαγές αυτές έχουν δημιουργήσει νέες ε, δυνατότητες, αλλά και νέα ευθύνη για την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία των πολιτών. Το 2007 ε, ξεκίνησε η ε, πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την δημιουργική και πολιτιστική οικονομία. Και στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες προοπτικές. Έχουμε εδώ την συνεργασία ανάμεσα στην δημιουργική οικονομία και άλλους ε, τομείς καθώς ε, και προσφορές δικτύωσης, ε, ακροάσεις με ανθρώπους από τους διάφορους τομείς, ετήσια παρακολούθηση σχετικά με την εξέλιξη του τομέα αυτού, οικονομικός διάλογος για την αντιμετώπιση της πειρατείας στο ίντερνετ, καθώς και ο διαγωνισμός για ε, νέα πιλωτικά προγράμματα είναι περαιτέρω μέτρα από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Ε, το U Institute ε, είναι ο νέος φορέας του Κέντρου Δεξιοτήτων και έχει ξεκινήσει τις εργασίες του το 2016 στο Βερολίνο. Έτσι υπάρχουν νέες προσφορές και Εργαζόμαστε ιδιαίτερα, ε, ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την επιστημονική ανάλυση και την ε, μετάδοση των γνώσεων. Θέλουμε ε, να προωθήσουμε την ε, καινοτομία και πέρα από αυτό έχουμε σχεδιάσει community management με πολλαπλασιαστές των τάσεων και ανθρώπους που θα εξετάσουν τις νέες τάσεις. η αρμοδιότητα για τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, στην Γερμανία ανήκει στα κρατήδια. Έτσι λοιπόν ε, παίζουν και αυτά σημαντικό ρόλο. Σχεδόν σε όλα τα κρατήδια ε, δίδονται υποτροφίες, ενισχύσεις και άλλα είδη οικονομικής υποστήριξης. Στο μεταξύ λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια δομή εντός των κρατηδίων και το Αμβούργο ε, είναι ιδιαίτερο παράδειγμα αυτό. Το 2010 η ε, δημιουργική εταιρεία του Αμβούργου ιδρύθηκε και αποτελεί αρμόδιο γραφείο και χώρο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης όλων των φορέων ε, στην ε, δημιουργική οικονομία. Υπάρχουν, ε, για παράδειγμα, βάσεις δεδομένων, διατίθενται ακίνητα, υπάρχουν σύστημα ενισχύσεων μέσω συμμετοχικής χρηματοδότησης, προγράμματα παροχής συμβουλών και κατάρτισης, δίδονται νομικές συμβουλές ε, και προσφορές μετεκπαίδευσης. Έτσι καλύπτουμε λίγο πολύ το συνολικό φάσμα. Ε, αρχικά η ενίσχυση ήταν χρονικά περιορισμένη, αλλά ε, η γερουσία του Αμβούργου αποφάσισε να συνεχίσει επαόριστον της εργασίας αυτής της εταιρείας. Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί το Αμβούργο υπόδειγμα όσον αφορά την πρωτοβουλία για τη δημιουργική οικονομία. Παρ' όλα αυτά έχουμε την ε, πρόκληση της διατομιακής συνεργασίας του γεωγραφικού κατακαιρματισμού και της ε, ανάγκης για κεφάλαια. Από τη μία συχνά ο τραπεζικός τομέας δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αναλύσει τις πρωτοβουλίες του τομέα αυτού. Από την άλλη ε, είναι τόσο μεγάλη η πολυμορφία και η πολιτική συνήθως ε, θέλει να ευνοήσει εξίσου όλους τους τομείς. Ε, στην πράξη, λοιπόν, ε, υπάρχουν ακόμα προβλήματα, αλλά ο στόχος μας ε, είναι να βελτιώσουμε τις δυνατότητες για καινοτόμες μικρές πολιτιστικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και για το τελικό σας σχόλιο, γιατί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η διαφορετική νοοτροπία που θα πρέπει να υπάρχει για τις πιστώσεις στην Ευρώπη είναι ένα από τα θέματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ε, κλείνει λοιπόν εδώ αυτό το πάνελ, το οποίο ε, είχε, είναι, ήταν η δεύτερη παρέμβαση αυτής της θεματικής ενότησης και πριν κλείσω θα ήθελα να ρωτήσω αν η Προεδρία ή αν η Επιτροπή θέλουν να απαντήσουν ή αν θέλουν να προσθέσουν κάτι, αν μπορούν να διευκρινίσουν κάτι. Παρακαλώ.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 Ευχαριστώ κύριε Ράχτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, γιατί πολλά από τα θέματα που αναφέρθηκαν σήμερα το απόγευμα είναι πολύ σημαντικά και ήταν πολύ πλούσιο αυτό το απόγευμα. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά σας. Ε, το να ζητάμε περισσότερα χρήματα είναι το εύκολο, αλλά δεν ξέρω αν είναι το πιο εύκολο να τα συζητάει κανείς με υπουργού οικονομικών. Προς το παρόν το πλαίσιο μέχρι το 2020 έχει καθοριστεί και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εντός του πλαισίου τι ε, ε, κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, να σας πω δύο λόγια. Προς το παρόν, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που συζητήθηκε και σήμερα το απόγευμα, ε, εξετάζουμε να δούμε ε, με τα χρήματα που έχουμε τι αξία μπορούμε να έχουμε. Και αυτό προσπαθούμε να εξετάσουμε. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε αυτές τις πτυχές βάσης στοιχείων και θα έχουμε στατιστικά στοιχεία από τη Eurostat σύντομα, τα οποία θα αφορούν περισσότερο την ε, πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο προς το παρόν, ήταν ανύπαρκτο αυτό, επομένως μπορεί έτσι να έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση. Δεν είναι όμως του παρόντος, ε, μπορεί να γίνει αργότερα. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο εξεργαζόμαστε είναι μια μελέτη για τις αλυσίδες αξίες ε, του δημιουργικού κλάδου, γιατί συχνά δεν ξέρουμε ποια είναι η σχέση μεταξύ πολιτισμού και καινοτόμων βιομηχανιών, τι είναι πολιτισμός, τι είναι καινοτόμο. Δεν είναι πάντα εύκολη αυτή η σύνδεση. Ε, με τον Κρίστιαν Έλλερ τις προάλλες ε, και πάντα αναφέρεται στη βιομηχανία της μόδας ο κύριος Έλλερ και λέει ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς της Ευρώπης. Είμαι βέβαιη μετά από αυτά που είπε και ο Γάλλος συνάδελφος σήμερα ε, είμαι βέβαιη ότι για τον ορισμό του αυτό δεν ξέρω αν είναι αυτό ο πολιτισμός, αλλά υπάρχουν ε, θέματα τα οποία αφορούν διάφορους τομείς, διότι αναφέρεται μόνο στους μεγάλους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα σας πω ονόματα, αλλά κάποιες από αυτές τους οίκους μόδας είναι γαλλικοί, επομένως θα ξέρετε περί ποιον αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο πρέπει να εξετάσουμε από άλλο πρίσμα και να δούμε όλα αυτά τα θέματα με πιο οριζόντιο τρόπο. Πρέπει βεβαίως ε, μέσω και της ψηφιακής αλλαγής να εξετάσουμε λίγο καλύτερα τι κάνουμε και θα είμαστε έτοιμοι μέχρι τον Ιανουάριο. Ένα άλλο θέμα που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα δίκτυο δημιουργικών κόμβων. Ε, αναφερόμαστε σε ε, οικοσυστήματα, θερμοκήπια, λέξεις οι οποίες είναι πολύ της μόδας αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τι υπάρχει και τι λειτουργεί αποτελεσματικά, διότι προς το παρόν ξεφυτρώνουν παντού αρκετές πρωτοβουλίες, πολλές από αυτές χρηματοδοτούνται από τη Δημιουργική Ευρώπη, κάποιες άλλες όχι, αλλά εν τέλει αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και δεν αφορά μόνο τους δημιουργικούς κόμβους, κάποιοι από εσάς αναφέρθηκαν στη δημιουργικότητα εν γέννη. Ε, πώς μαθαίνουμε τη δημιουργικότητα, αυτά είναι από τα βασικά ζητήματα και πότε πότε κάνω το εξής. Ε, Ξέρετε ότι ο εγκέφαλο λειτουργεί και από την αριστερή και από τη δεξιά πλευρά. Προσπαθώ να τα διαχωρίσω λοιπόν, δεν είναι πάντα εύκολο. Και προσπαθώ να σκεφτώ και στα εκπαιδευτικά συστήματα που μπορούμε να τα εντάξουμε αυτά. Πολύ συχνά αναφερόμαστε στα θέματα αυτά μόνο από τη δημιουργική σκοπιά ή είσαι δημιουργικό ή δεν είσαι, αλλά αυτό που προσπαθώ να δω τώρα είναι πώς μπορούμε να βρούμε τρόπους και στον εκπαιδευτικό κόσμο ε, να ε, καταφέρουμε να έχουμε πιο δημιουργικά παιδιά. Ε, η δική μου γενιά νομίζω δεν διδάχθηκε να είναι δημιουργική. Αυτοί που διδάχτηκαν ήταν καλά και ωραία, αλλά για τους υπόλοιπους ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν ήταν τμήμα της ύλη του σχολείου αυτό. Δεν ήταν έπρεπε να είσαι αυτό το οποίο σου εδίδασκε ο δάσκαλος. Ναι μεν, αλλά τώρα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους ώστε οι νέοι, τα νέα παιδιά ε, να ε, έχουν το περιθώριο να είναι δημιουργικά. Αυτό λοιπόν αφορά και την εκπαιδευτική σκοπιά. Πρέπει να έχουμε λοιπόν παιδεία, πολιτισμό, καινοτομία από κοινού. Όλα αυτά τα θέματα ε, ενώνονται και πρέπει να τα εξετάζουμε ως σύνολο. Αναφέρθηκε κάποιος στο crowdfunding. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ε, και την καινοτομία στον πολιτισμό με διαφορετικό τρόπο. Ε, Μία συζήτηση που κάναμε όταν έγινε το πολιτισμικό φόρουμ πριν από κάποιους μήνες είναι ότι δεν μπορούμε να βρισκόμαστε σε ένα σύστημα στο οποίο θα ζητούμε συνέχεια περισσότερα χρήματα. Κάποια στιγμή ε, τα κονδύλια αυτά είναι περιορισμένα. Η δική μου η έκκληση λοιπόν είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά αυτά τα χρήματα. Στο σημερινό κόσμο και στον κόσμο των παιδιών μας υπάρχουν πολιτιστικές ανταλλαγές, υπάρχει ε, μια κουλτούρα ανταλλαγής και συμμετοχής και νομίζω ότι ε, ο κόσμος που γνώριζα εγώ όταν ήμουν στα 20 δεν είναι ο ίδιος με το σημερινό κόσμο. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ πιο δημιουργικά τι ε, χρειάζονται οι δικοί μας οι νέοι ε, και τι ζητούν. Και όταν δω τι βλέπουν στο YouTube ή οπουδήποτε αλλού, δεν είναι αυτό που βλέπουμε κι εμείς. Και υπάρχουν τρόποι ε, να, οι τρόποι μάλλον με τους οποίους διδάσκονται οι ίδιοι τον πολιτισμό είναι τελείως διαφορετικοί από τον τρόπο με τον οποίο διδασκόμασταν εμείς. Επομένως πρέπει οι νέοι ε, να συμμετέχουν πολύ περισσότερο από όσο καταφέραμε μέχρι τώρα και κυρία Πρόεδρε αν μου επιτρέπετε είναι κάτι το οποίο ε, μου λείπει από το σημερινό ε, απόγευμα και είναι κάτι το οποίο θα ήταν τελείως ξαφνικό και είναι πολύ σημαντικό και ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ότι οι νέοι δεν είναι μαζί μας. Είναι κάπου αλλού και επομένως πρέπει να τους πάρουμε μαζί μας. Γι' αυτό τώρα ε, εργαζόμαστε και για το δίκτυο νέων δημιουργικών επιχειρηματιών. Ο όρος ε, entrepreneur επιχειρηματίας είναι πολύ της μόδας και αυτός, αλλά πρέπει να κάνουμε μια σχέση μεταξύ δημιουργίας και επιχειρηματικότητας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μια τελευταία φράση που είναι μια έκκληση. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018. Να ευχαριστήσω και πάλι την Πρόεδρο, την κυρία Κώστα και όλους εκείνους που μας βοήθησαν να έχουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος. Ε, όλοι συμμετέχουμε μαζί σε αυτό και πρέπει λοιπόν να ε, αποτελέσει επιτυχία. Δεν είναι θέμα χρημάτων, σίγουρα χρειάζομαστε χρήματα, αλλά ε, είναι και θέμα καινοτομία. Να αποδείξουμε ότι μπορούμε από κοινού να εξηγήσουμε ε, την Ευρώπη με τον καλύτερο πολιτιστικό τρόπο προς τους πολίτες μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέου τρόπου λειτουργία, νέου τρόπου επικοινωνία, νέου τρόπου για να πείσουμε τους νέου ανθρώπου να συμμετέχουν. Ε, Τις προάλλες ήμουνα μπροστά από 5.000 ε, προσκόπους. Πώς μπορούμε να τους πείσουμε λοιπόν να συμμετέχουν και να συμμετέχουν στον πολιτισμό. Διότι ο τρόπος που εξετάζουμε και βλέπουμε εμείς τον πολιτισμό δεν είναι ο ίδιος τρόπος που τον εξετάζουν και τον βλέπουν αυτοί. Πρέπει λοιπόν να τα έχουμε αυτά από κοινού, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και τα δύο και προς το παρόν αυτό για μένα είναι ερωτηματικό ακόμα. Ε, ευπρόσδεκτη λοιπόν ε, ιδέα, χρειάζομαι πολύ καλές ιδέες. Ε, το 2018 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε. Πώς μπορούμε να προβάλλουμε περισσότερο τον πολιτισμό μας. Με αυτή τη μικρή ερώτηση λοιπόν, Αστείευομαι βεβαίω. Πολύ δημιουργική η Γενική Διευθύντρια. Μα αφήνει το ερώτημα να εωρείτε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ένα πολύ μικρό, πολύ μικρό παράδειγμα. Σήμερα εμεί βραβεύσαμε τρει νέου οι οποίοι κέρδισαν το βραβείο Καρλομάγνο για του νέου. Ένα εξ αυτών είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων που έφτιαξαν ένα βιντεοπαιχνίδι για τον Καρλομάγνο. Και είπα, γιατί εμεί είμαστε δημιουργικοί αυτή τη στιγμή, μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα, γιατί στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού έτου ή και νωρίτερα να μην ξεκινήσει μία πρόσκληση διαγωνισμού για ε, εφαρμογέ, τι οποίε θα φτιάξουν οι νέοι που θα δημιουργούν και θα διηγούνται την Ευρώπη. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι το σκέφτηκαν αυτό μαθητέ Λυκείου από τον πύργο και ε, έφτιαξαν ένα βίντεο για τον Καρλομάγνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ε, πραγματικά ε, συμφωνώ και εγώ, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε την κατάλληλη γλώσσα να μιλήσουμε τους, στους νέους. Πρέπει να βρούμε πώς μπορούμε να συνομιλούμε. είχαμε και μια έκθεση για το πώς να ετοιμάσουμε την Ευρώπη σχολείο. Ε, ο συνάδελφος Ντράγκη παρουσίασε την έκθεση και ο συνάδελφος Ντράγκη έχει μια ιδιαίτερη ιστορία διότι ε, είναι μέλος της κοινότητας των Ρωμά. Ε, μας εξήγησε λοιπόν πόσο πολύ ενδιαφέρον είχε για αυτόν και για, λόγω της προσωπικής του ιστορία να φτιάξει μια Ευρώπη ε, από ένα τελείως διαφορετικό οπτικό πρίσμα. Εάν συμφωνείτε τώρα θα ε, περάσω απευθείας στο επόμενο πάνελ γιατί περνάει ο χρόνος για... την συμμετοχή των πολιτών στον πολιτισμό. Είμαστε πολύ κοντά λοιπόν σε αυτή την πρόκληση ε, για τον πολιτισμό. Η κυρία Κριστίνα Νταμιλάνο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πολιτιστική Οργάνωση και Διαχείριση θα κάνει την παρουσίαση. Ξέρω ότι ζητά πολύ ευγενικά ο συνάδελφο Διακόνου, τον οποίο αναφέραμε προηγουμένω γιατί είναι εισηγητή για το Ευρωπαϊκό Έτο για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ε, να μιλήσει πρώτος ε, γιατί πρέπει να βρίσκεται σε κάποια άλλη υποχρέωση. Δεν ξέρω αν μπορεί να μιλήσει πρώτα η προγνώμονάς μας. Κύριε Διακόνου, πόσο χρόνο έχετε. Να δώσω το λόγο στην εμπειρογνώμονα πρώτα και μετά σε εσά. Τέλεια. Ωραία. Καλύτερα έτσι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσω Ιταλικά ώστε να είμαι βέβαιη ότι θα σεβαστώ και τους χρόνους. Έτσι μπορώ να είμαι και λίγο πιο συνοπτική αν χρησιμοποιώ τη γλώσσα μου. Ε, έχω κάποιες διαφάνειες για σας στις οποίες διαφάνειες φυσικά ε, έχω χρησιμοποιήσει την αγγλική γλώσσα και θα χρησιμοποιώ και την αγγλική ορολογία όταν θα αναφέρομαι στο audience engagement και στο audience development, ε, διότι ε, ορισμένες φορές χανόμαστε στην μετάφραση κάποιων όρων και είναι πολύ περίπλοκα αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε όλοι μαζί την ίδια αγγλική ορολογία. Για να μιλήσουμε λοιπόν για engagement, για συμμετοχή των πολιτών στην, στον πολιτισμό, πρέπει να ε, αναρωτηθούμε το εξή καταρχάς γιατί το κάνουμε. Γιατί λοιπόν αναφερόμαστε σε ε, δέσμευση, σε συμμετοχή, σε engagement. Ε, γιατί τα στοιχεία μας αποδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα ελάχιστοι άνθρωποι στην Ευρώπη συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από την εξή προπόθεση, ότι όλη η διαδικασία εκδημοκρατισμού του πολιτισμού που έγινε την τελευταία πεντηκονταετία δεν έχει ε, επιτύχει πλήρω του στόχου τη. Σαφώ η υποστήριξη τη πρόσβαση και τη συμμετοχή αποτελούν προτεραιότητα στι ε, πολιτιστικέ πολιτικέ ε, τη Ευρώπη και επομένω η συμμετοχή και η ανάπτυξη του κοινού είναι δύο από του πυλώνε για την προώθηση των πολιτισμικών αξιών και τη ενεργού ηθαγένεια. Τι εννοούμε με τον όρο audience engagement. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένας όρος ο οποίος ε, αφορά τη διάσταση της συμμετοχής, αλλά είναι ένα σύνολο διαδικασιών, δράσεων και συμπεριφορών και κυρίως πρόκειται για κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με την ε, ιδέα της ε, ανάπτυξης ε, του κοινού, του audience development. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από τον ορισμό του audience development όπως δίνεται στην Δημιουργική Ευρώπη για παράδειγμα. Το audience development είναι μια διαδικασία στρατηγική, δυναμική και διαδραστική η οποία επιτρέπει να είναι προσβάσιμος ο πολιτισμός που σημαίνει ότι ε, βοηθά στη συμμετοχή των πολιτών και των κοινοτήτων και το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία της εξέλιξης με τρεις τρόπους. Καταρχάς, ή προσπαθούμε να διευρύνουμε σε ποσοτικούς όρους ε, του παραδοσιακού κοινού ή να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ αυτού του παραδοσιακού κοινού, σε μια κάθετη δηλαδή σχέση, ή με ένα τρίτο τρόπο που είναι η διαφοροποίηση του κοινού. Δηλαδή προσπαθώντας να επιτύχουμε ε, και την πρόσβαση σε κοινό που δεν είναι το παραδοσιακό μας κοινό. Γιατί επικεντρώθηκα λοιπόν σε αυτούς τους ορισμούς. Αυτή τη στιγμή συμμετέχω σε μια ομάδα εργασίας η οποία... Ε, εκπονεί μία μελέτη που ε, ζήτησε η Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού, που κάνει μία μελέτη για την ανάπτυξη του κοινού για το πώς μπορεί το κοινό να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτιστικών οργανώσεων. Πώς μπορούν λοιπόν οι πολιτιστικές οργανώσεις να βάλουν το κοινό στο επίκεντρο ε, των προσπαθειών τους. Πρόσκειται λοιπόν για μια δουλειά η οποία βασίζεται κυρίως σε βιβλιογραφική έρευνα, αλλά κυρίως ε, μέσω περιπτωσιολογικών μελετών. Ε, αναζητήσαμε στην Ευρώπη περιπτωσιολογικές μελέτες μουσείων, βιβλιοθηκών που ασχολούνται με προσέγγιση του κοινού. Επιλέξαμε 30, όπως βλέπετε από το χάρτη, από τις πάνω από 80 προτάσεις που έχουμε λάβει, 30 από περίπου ε, όλη την Ευρώπη. Βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάλυσης αυτών των περιπτώσεων. Ε, προς το τέλος του έτους θα έχουμε τα αποτελέσματα και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω μεταξύ είναι ότι έχουμε ε, διαπιστώσει κάποιες τάσεις και μέσω της βιβλιογραφίας και μέσω της ανάλυσης των περιπτωσιολογικών μελετών. Καταρχάς, υπάρχει μια αλλαγή όσον αφορά το, την ορολογία που χρησιμοποιείται, των συγκεκριμένων όρων. Από πρόσβαση στον πολιτισμό πάμε στον όρο audience development και ε, αυτό γίνεται συνειδητά από τον έναν όρο στον άλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις το audience development αφορά ε, διαστερεότητες που αφορούν περισσότερο την κοινωνική ένταξη, επομένως πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μετρήσουμε την κοινωνική επιρροή ε, της πολιτιστικής δομής ε, προϋποθέτει οργανωτική ε, αλλαγή και αλλαγή ηγεσία. και φυσικά ε, θέματα που αφορούν τη συμμετοχή και την δέσμευση και υπάρχει και το όλο θέμα της αλλαγής σε ψηφιακό επίπεδο. Αυτά τα αποτελέσματα θα δείτε στο τέλος του έτους. Θα ολοκληρώσω με δύο παρατηρήσεις και μία τελευταία υποσημείωση. Καταρχάς, δεν μπορούμε να έχουμε εργασία για τα θέματα αυτά αν δεν υπάρχει και μία προσπάθεια σε εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες θα αποτελούν κίνητρο και θα ε, ευνοούν την, το ενδιαφέρον για την τέχνη το, και τον πολιτισμό. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τα μουσεία και τις βιβλιοθήκες να καλύψουν ένα εκπαιδευτικό κενό, το οποίο αναφέρθηκε άλλωστε σήμερα. Η άλλη πτυχή είναι πολύ συχνά ε, το γεγονός ότι τα ε, πολιτιστικά ιδρύματα μετά την εφηβεία χάνουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να έχουμε ε, διαβίου μάθηση και για τους ενήλικες σε μη τυπική διαδικασία. Και ολοκληρώνω για να σας πω επίσης ότι θεωρώ ότι όλα αυτά δεν έχουν ε, ε, νόημα, το λέω βεβαίως ως ερευνήτρια, όχι ως πολιτικός, εάν δεν έχουμε ε, τους τέσσερις πυλώνες της βιωσιμότητας. Όχι μόνο οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, αλλά και πολιτιστική βιωσιμότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία σύνοψη και με πολύ ενδιαφέρον θα διαβάσουμε βεβαίως και την έρευνά σας. Ε, ελπίζω ότι όταν θα είναι διαθέσιμη, το ζητώ και από την κυρία Ρέχτερ, να τη διανύμουμε γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Αυτή η συζήτηση λοιπόν για το engagement και το development είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, διότι πρέπει να ε, είμαστε και πιο δραστήριοι. Ωραία, να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Διακόνου ο οποίος είναι εισηγητής ε, της έκθεσης προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ε, πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, μια πολύ σημαντική έκθεση βάσει της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε πέρσι και τώρα είναι εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018. Παρακαλώ κύριε Διακόνου. Ε, ε, δηλαδή Συγγνώμη, ο κύριος Διακόνο είναι εκπρόσωπος των Φιλελευθέρων και είναι ένας εκ τους αντιπροέδρων της Επιτροπής Πολιτισμού. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να πάρω τη σκητάλη από την προηγούμενη με ομιλήτρια για να πω ότι καταλάβαμε κάτι πολύ σημαντικό. Η διαφορά μεταξύ των ανθρωπίνων όντων και των ρομπότ είναι η κουλτούρα, ο πολιτισμός και γι' αυτό οι άνθρωποι είναι ανώτεροι των ρομπότ και γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό. Δεν είναι χρήσιμο να έχουμε άψογη και τέλεια οικονομική αποτελεσματικότητα χωρίς όμως πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά. Το ανήκει σε μια κουλτούρα, σε μια ιστορία, σε ένα πολιτισμό είναι αυτό το οποίο καθιστά το ανθρώπινο όν ανώτερο των λοιπόν ειδών. Σε κάθε περίπτωση ε, πολύ γρήγορα θα ολοκληρώσουμε την ε, σχετική έκθεση για τα θέματα πολιτισμού. Θα είναι έτοιμη σε δύο-τρεις εβδομάδες και θα προχωρήσει η έκθεση αυτή βάσει της διαδικασίας του κάθε κατεπήγοντος γιατί έχει νομοθετικό ε, αποτέλεσμα. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και έχουμε και την πολύ μεγάλη τύχη έχουμε και την πολύ μεγάλη τύχη η σημερινή μας προσκεκλημένη να είναι ακριβώς οι άνθρωποι που χρειάζεται έτσι ώστε να έχει συνέχεια αυτή η έκθεση στο μέλλον, να μπορέσει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμοστεί σωστά. Μιλώ για την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και αυτή η έκθεση θα έχει αξία μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε βασιστεί στη συνεισφορά των κρατών μελών και βεβαίως των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Παρ' όλα αυτά, βασικό στόχος αυτού του κειμένου είναι ο εξής. Ο τρόπος με τον οποίο η κουλτούρα και η ιστορία μας μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα. Έχουμε κοινή ιστορία Και αυτό το αποτέλεσμα ελπίζουμε να έχουμε με το ευρωπαϊκό έτος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Να τονίσουμε ότι είμαστε μαζί, ε, η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει σε όλους μας και τη μοιραζόμαστε από κοινού όλοι μας. Και αυτά θα ήθελα να πω, ε, καταρχάς προσπαθώντας να προσεγγίσω ένα πρόβλημα που έχει εξαπλωθεί στην ευρωπαϊκή επικράτεια και αναφέρομαι στους εθνικισμούς, τους κατατόπους, ε, τους, τους οποίους πραγματικά δεν χρειαζόμαστε. Είναι ένα φαινόμενο που απαντάται σε πολλά Το 2017 θα είναι το έτος προετοιμασίας του έτους 2018 και σε επίπεδο προϋπολογισμού και σε επίπεδο δημοσιονομικό. Επομένως, η σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι απολύτως απαραίτητη, διότι χρειαζόμαστε τη δική σας στήριξη, χρειαζόμαστε όλους εσάς. Αυτή η χρονιά λοιπόν θα είναι επιτυχία μόνο εάν η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, οι τοπικές περιφερειακές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια σύσσωμα, σύσσωμοι όλοι αυτοί οι φορείς κάνουν αυτή την προσπάθεια να ε, διαδώσουν όλα αυτά που μας ενώνουν, όλα αυτά που αποτελούν την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά. Η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί το αργότερο το Δεκέμβριο και θα συνεχίσουμε την επικοινωνία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σε κάθε περίπτωση δράτω με τις ευκαιρίες για να χαιρετήσω τους δύο Ρουμάνους συναδέλφους, ε, προέδρους των αντιστοίχων Επιτροπών Πολιτισμού των δύο τμήματων του Ρουμανικού Κοινοβουλίου και χαίρομαι διότι βλέπω και τους λοιπούς συναδέλφους εδώ. Κοινή είναι η στόχη μας και ελπίζω ότι θα έχουμε επιτυχία. Θέλησα όλα αυτά να σας τα πω τώρα για να γνωρίζετε ότι το, 2018 θα έρθει, θα είναι το έτος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να δείξει το δικό της κομματάκι, αυτό που αυτή έχει ε, καλύτερο. Και αυτό εμεί το ονομάζουμε εκδημοκρατισμό της κουλτούρας και του πολιτισμού. Δεν υπάρχει μία κουλτούρα μίας χώρας που είναι πιο σημαντική από αυτή ε, της άλλης ε, χώρας. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος συνεργασίας, ενεργής, δραστικής και ελπίζω όλα αυτά με να στεφθούν με επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί όντω έγινε μια συζήτηση για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμού ε, που, πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι ένα πολύ καλό ε, σημείο κίνησης. Να υπενθυμίσω ότι το 2017 θα είναι έτος προετοιμασίας και πολύ μεγάλη συμμετοχή των κρατών μελών. Επομένω, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας χώρος διακυβέρνησης ε, όπου μπορούν φυσικά να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια για να συμμετέχουν όλες οι δομές ενώσεις, ε, το ε, περιφερειακό επίπεδο, το τοπικό επίπεδο. Κάνουμε αυτή την έκκληση γιατί πρέπει να αντιληφθούμε όλα αυτά τα θέματα. Επίσης πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση της κληρονομιάς. Όχι μόνο κάθε χώρα να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, πρέπει να υπάρχει και μια πιο ευρωπαϊκή διάσταση. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το γνωρίζει ήδη άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί το είπαμε ε, ήδη σε αρκετές περιπτώσεις, εμείς εγκρίναμε ευτυχώς ε, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, μετά από την Επιτροπή Πολιτισμού να ε, υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια και το 2017 φυσικά και το 2018 μέσω μιας ανεξάρτητης γραμμής προϋπολογισμού και όχι να παίρνουμε πόρους από ε, προγράμματα όπως το Δημιουργική Ευρώπη που έχουν ήδη περικοπεί ε, αρκετά. Ε, κάνω έκκληση λοιπόν και προς τη Σλοβακική Προεδρία και προς όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξουν το θέμα αυτό. Η πίεση των κρατών μελών και των εθνικών κοινοβουλίων θα ήταν εξαιρετική βεβαίω γιατί θα βοηθούσαν για το στοιχείο αυτό το οποίο θα είχε θετικές συνέπειες βεβαίω και για το δικό σας το ρόλο. Να δώσουμε αμέσω το λόγο στον Dragon Matic για την παρουσίασή του. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Σλοβενίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Σλοβενία παραδοσιακά έχει πολιτιστικό προσανατολισμό στο χάρτη μας. Βλέπετε ότι επί ε, αιώνες ε, έμεναν, ε, ζούσαν σε διάφορες ενότητες, διάφορες ενώσεις. Παρ' όλα αυτά η κοινή γλώσσα και ο κοινός πολιτισμός τους ενώνει. Η εθνική ταυτότητα έχει αντικαταστήσει το ρόλο του κλασικού κράτους έθνους χαρακτηριστικό είναι ότι στα παλιά μας νομίσματα πριν το ευρώ είχαμε καλλιτέχνες ε, ως μορφές ε, πάνω, επιστήμονες, ε, ζωγράφους, συγγραφείς, μουσικούς, όχι όμως πολιτικούς ή ήρωες του πολέμου. Η Σλοβενία επίσης είναι μοναδική στο ότι έχει ειδική πολιτιστική αργία ε, και έχουμε επίσης ε, την 8η ε, Φεβρουαρίου που είναι η λεγόμενη ημέρα Πρεσερέν. Επίσης έχουμε την ημέρα πολιτισμού της 3 Δεκεμβρίου που είναι τα γενέθλια του ε, Σλοβαίνου ποιητή Φρανς Πρεσερέν. Η Σλοβενία έχει πάνω από 4.900 ε, συλλόγους ε, ερασιτεχνών με σχεδόν 100.000 ε, μέλη. Επίσης, κατέχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ όσον αφορά τον αριθμό νέων βιβλίων που εκδίδονται κατά κεφαλήν. Οι περισσότεροι ε, Σλοβαίνοι, μάλλον κατά μέσο όρο, ε, επισκέπτονται τέσσερις φορές ε, τον χρόνο, συγγνώμη, 20 φορές τον χρόνο δημόσια βιβλιοθήκη. Δεν είναι πολύ εύκολο το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την συμμετοχή των πολιτών. Θα μπορούσαμε να διεισδύσουμε σε τομείς όπου δεν έχουμε διεισδύσει μέχρι τώρα, τον κοινωνικό, το περιβάλλον κλπ να χρηματοδοτήσουμε δηλαδή και τέτοια προγράμματα. Επίσης, θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε το ε, σύστημα ε, ε, πολιτιστικού πολιτισμού πολιτιστικής πολιτικής και θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα πρέπει να αναφέρουμε το ρόλο που παίζουν αυτές οι οργανώσεις στον τομέα του πολιτισμού, διότι αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα είναι πιο δημοκρατική, δημοκρατικές οι οργανώσεις αυτές και μπορούν να έρθουν πιο εύκολα σε επαφή με διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Για την προώθηση του, της συμμετοχής των πολιτών στον πολιτισμό, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους ε, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σλοβενία έχει υποβάλει πρόταση που συνδυάζει δύο πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την συμμετοχή νέων ε, στον πολιτισμό και το συνδυάζει με την ε, κινητικότητα προτάθηκε όλοι οι 18χρονοι να έχουν δωρεάν είσοδο σε πολιτιστικά ιδρύματα. Αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με το δώρο ενός εισιτηρίου Interrail σε κάθε νέο που συμπληρώνει τα 18 του χρόνια. Θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την πρόταση αυτή σε κάθε 18χρονο που ταξιδεύει στην Ευρώπη για να δει τις ομορφιές της Ευρώπης θα πρέπει να δίνουμε και την δυνατότητα να ε, επισκέφτεται πολιτιστικούς χώρους δωρεάν. Αυτό θα μας επέτρεπε να ενισχύσουμε την ε, πολιτιστική μας συνείδηση. Έτσι θα μπορούσαμε επίσης να πετύχουμε καλύτερα τους κοινούς μας στόχους. Εάν οι νέοι αγαπήσουν τον πολιτισμό τους, θα συνεχίσουν να ασχολούνται με αυτόν, ε, μέχρι τη γύρανσή τους. Ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Φλάβια Πίκολη Ναρτέλη, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού της ε, Βουλής των ε, Αντιπροσωπών της Ιταλίας. Καλησπέρα κυρία Πρόεδρε. Ε, στους συναδέλφους ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων και στους ε, συμμετέχοντες σε αυτή τη συνάντηση. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις προκλήσεις στον πολιτισμό και στη δημιουργικότητα και ακούσαμε μεγάλο ενδιαφέρον τους συναδέλφους από τις άλλες επιτροπές συνειδητοποιούμε όλοι ότι η προώθηση αυτών των τομέων αποτελεί κίνητρο για τα επιχειρηματικά συστήματα με θετικές εξελίξεις ε, στην ανάπτυξη των περιοχών μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο πολιτισμός και το μέλλον είναι ε, ένα αναπόσπαστο Γι' αυτό ακριβώ ε, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω του συναδέλφους από την Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πρόεδρο και την κυρία Κώστα που έδωσαν μεγάλη ε, μάχη προκειμένου να συμπεριληφθεί η δημιουργική Ευρώπη στο Ευρώπη 2020. Θεωρώ ότι το στίχημα κερδίθηκε και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Επίση, θα θέλαμε να υποστηρίξουμε την πρόταση το 2018 να είναι το Ευρωπαϊκό Έτο πολιτιστική κληρονομιά. Νομίζω ότι και επ' αυτού είναι πολύ χρήσιμο και πολύ πολύ σημαντικό να επενδύσουμε όλοι. Τα τελευταία δύο χρόνια στην Ιταλία είχαμε μια σειρά από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για την πρόθεση του πολιτισμού και λόγω της τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς ε, που διαθέτει. Σε γενικές γραμμές ε, η κατάσταση προβλέψεων ε, του Υπουργείου Πολιτισμού έχει ένα πολύ σημαντικό αριθμό, ε, πάνω από 3,7% αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και προσπαθεί να κάνει μια αναδιοργάνωση του συστήματος των μουσείων της Ιταλίας. Στο μεταξύ, το, Υπουργό, το Υπουργείο Παιδείας, ε, Πανεπιστημίων και Έρευνας ε, επένδυσε πάρα πολλά κονδύλια στα σχολεία για την κατάρτιση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέα εναλλαγή ε, ε, εναλλαγής εργασία, προσπαθώντα να συνδυάσουν τον κόσμο του σχολείου, τον κόσμο του πολιτισμού και βεβαίω τον κόσμο τη καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα, στο νόμο σταθερότητα για το 2016 υπήρξαν πάρα πολλέ παρεμβάσει, μεταξύ των οποίων θα ήθελα να αναφέρω, όπω και υπενθύμησε και ο προηγούμενο συνάδελφο ε, την κάρτα πολιτισμού για του νέου που συμπληρώνουν τα 18 τους για να ξοδέψουν για πολιτιστικά αγαθά, όπως για παράδειγμα αγορά βιβλίων κτλ. Και επίσης ένα τριετές ταμείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ε, με 400 εκατομμύρια ευρώ για την ε, καταπολέμηση της πολιτιστικής ένδυας ε, και θέλουμε να επενδύσουμε σε παιδιά διότι μόνο μέσω αυτής της επένδυσης στον πολιτισμό μπορούμε να ανακτήσουμε τα όσα έχουμε χάσει. Επενδύοντας λοιπόν στον κόσμο του βιβλίου και του πολιτισμού εν γέννη, στο, στη Βουλή ένα σχέδιο για την προώθηση της ανάγνωσης, ένα σχέδιο το οποίο θα βοηθήσει βιβλιοθήκες, ε, ε, βιβλιοπολία και αναγνώστες για να διευρύνουμε το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο από το 2014 υπάρχει και ένα art bonus ε, το οποίο θα ήθελα να υπενθυμίσω. Ένα σύστημα πρημοδότησης ε, το οποίο αντιστοιχεί στο 75% για δωρεές για πολιτιστικά αγαθά το οποίο αποτελεί επιτυχία στην εφαρμογή του και ουσιαστικά ε, βοηθά ε, στην δημόσια και ιδιωτική σύμπραξη για την αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όσον αφορά τη δημιουργική βιομηχανία, είμαι βέβαιη ότι η δημιουργική βιομηχανία μπορεί να διαχέει ιδέες και να απευθυνθεί σε διαφορετικό κοινό και αυτό φυσικά βοηθά στην ποικιλομορφία της χώρας. Χάρη στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ε, θα έχουμε σημαντικούς πόρους για έργα στον τομέα του πολιτισμού, στον οπτικοακουστικό τομέα και επίσης θα θέλαμε να αυξηθούν αυτό ακριβώ ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει το αίτημα της επαναχρηματοδότηση, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί. Επιπλέον, Θεωρούμε ότι το Scoping Paper του 2018-2020, το οποίο περιορίζει το ε, τα σημεία παρέμβασης θεωρεί ότι ο πολιτισμός είναι μία από τις τρεις μακροπεριοχές για το πρόγραμμα εργασίας 2018-2020. Αυτές τις εβδομάδες στην Επιτροπή Πολιτισμού της Βουλής συζητούμε μία πρόταση νόμου για να υποστηρίξουμε τις δημιουργικές βιομηχανίες από την αρχή τους, ε, χρησιμοποιώντας την εμπειρία των νεοφυών επιχειρήσεων στο τεχνολογικό τομέα, που ε, έχουν ε, μέσω διατάγματος ε, ανάπτυξη 2.0 καλύτερο ευνοϊκό περιβάλλον και συγκεκριμένη ρύθμιση ad hoc για να προωθήσουμε και κάποιες προτάσεις και να απαντήσω στο τι ακριβώς κάνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια για να υποστηρίξουν τις τομείς αυτούς. Έχουμε περίπου 6.000 startup επιχειρήσεις στην Ιταλία με αύξηση πάνω από 50% των ανθρώπων που συμμετέχουν, υπαλλήλων και εταίρων. Όσον αφορά τις συνέπειες της ε, τεχνολογικής καινοτομίας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, η ψηφιακή πρόκληση μπορεί να συνεισφέρει στο πλήρες δικαίωμα πρόσβασης και αξιοποίησης των πολιτιστικών αγαθών, ε, βελτιώνοντας τη γνώση που πρέπει να βρίσκεται στη βάση της παγκόσμιας οικονομίας. Προωθούμε λοιπόν την ψηφιοποίηση της κληρονομιάς μας, κυρίως στο πλαίσιο των στρατηγικών για μια ενιαία ψηφιακή αγορά, και αυτή τη στιγμή στη Γερουσία ε, διαβάστηκε η πρόταση οδηγίες Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την παροχή οπτικοακουστικών μέσων που παρεμβαίνει σε συγκεκριμένα προφίλ που δεν έχουμε ξανακούσει όσον αφορά τους παρόχους πλατφόρμας για την ανταλλαγή βίντεο ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την προστασία των ανηλίκων και όλων των χρηστών. Τελευταίο σημείο, αυτή τη στιγμή ε, στη Βουλή των Αντιπροσώπων ε, εγκρίνεται το σχέδιο μεταρρύθμισης ε, του οπτικοακουστικού τομέα και του τομέα του κινηματογράφου. Θα το εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Επιτροπή Πολιτισμού θα τα εξετάσει με τη δέουσα προσοχή. Ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα όσα έγιναν. Και τώρα έχουμε τον κύριο Γεώργη Κασεβερίν, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης της ε, Γερουσίας της Ρουμανίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί οργανωτές αυτής της συνεδρίασης, χαίρομαι γιατί μπορώ να σας απευθύνω χαιρετισμούς από τη γεωρουσία της ε, Ρουμανίας και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει για το ότι αυτή η Επιτροπή είναι πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Ευρωβουλευτών και μελών Εθνικών Κοινοβουλίου μπορούν ο τομέας ο πολιτισμικός και ο πολιτιστικός να συμβάλλει ιδιαιτέρως στην οικονομία της χώρας. Η προώθηση αυτών των κλάδων θα δώσει μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα μας. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Θα ε, προσελκύσουμε επενδύσεις διότι ε, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία και έχουμε εξελίξει σε κοινωνικό επίπεδο ε, στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό. Σίγουρα οι υποδομές είναι ανεπαρκείς, σίγουρα ε, είναι λυπής η κατάρτιση των επαγγελματιών και σίγουρα υπάρχει αβεβαιότητα στους εργαζόμενους γιατί την εποχιακή η εργασία πολύ συχνά και δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Όλα αυτά θέλουμε να τα ανατρέψουμε. Ε, έχει συζητηθεί ιδιαίτερο το θέμα αυτό και έχει μελετηθεί σε πολλές μελέτες. Υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Στη Ρουμανία έχουμε στρατηγική για την περίοδο 2016-2020, προγραμματικό πλαίσιο δηλαδή, και θεωρούμε ότι για να εμπλέξουμε περισσότερο τους πολίτες στην πολιτιστική ζωή, τότε πρέπει να ενισχύσουμε την πρόσβαση στις υποδομές πολιτισμού. Και όταν παράγεται και καταναλώνεται πολιτισμός από τους πολίτες, κουλτούρα και κυρίως από τους νέους, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις νέες τεχνολογίες και τα νέα μέσα επικοινωνίας που περιέχουν και μεγάλες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Η δημιουργία δικτύων και πλατφόρμας διαδικτυακής είναι κάτι το, πολύ, ε, το πολλά υποσχόμενο. Ε, θέλω να ευχαριστήσω το, το προσωπικό του γραφείου που μου ετοίμασε την ομιλία, αλλά δεν θα μιλήσω πια διαβάζοντας. Ε, θέλω να φύγω από το κείμενο και να μιλήσω για θέματα που παραγνωρίζουμε πολύ συχνά. Μιλούμε για τον τομέα της δημιουργίας και συνέχεια λέμε ότι πρέπει να επιλέξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μελη ε, στη διανομή του προϊόντος της κουλτούρας και του πολιτισμού. Καλώς και σωστά. Ωστόσο, η δημιουργία είναι υποκειμενικό πράγμα ε, και μπορεί να συμφωνούμε ή μπορεί να μην συμφωνούμε. Το σημαντικό είναι η έμπνευση του δημιουργού και η ευφυΐα του, το πνεύμα το καλλιτεχνικό. Εάν καταφέρουμε αυτό να προωθήσουμε, θα είναι αυτό πολύ επιτυχές. Δηλαδή, να μην καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα ε, συνεταιρίζεστε μια κουλτούρα βιομηχανική και μαζικής παραγωγής ε, προπολιτισμού γιατί έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να παραγνωρίσουμε ε, την καλλιτεχνική ιδιαιτερότητα. Τα μεγάλα έργα του ευρωπαϊκού πολιτισμού δημιουργήθηκαν από άτομα που κατάφεραν να επιβληθούν, κατάφεραν, τους επετράπη να δημιουργήσουν. Εάν ε, κάνουμε και μια αναδρομή ιστορική, η Αθήνα του Περικλή, η Φλωρεντία, ε, ε, τους, την οικογένεια των Μεδίκων, είναι χώροι πολιτισμού που κατέστησαν τέτοιοι γιατί τους επετράπη από τους πολιτικούς ηθήνοντες της εποχής. Θα πρέπει λοιπόν να καλλιεργήσουμε την οτροπία αυτή να, μια νοοτροπία στην οποία τα άτομα να μπορούν να λειτουργήσουν και να δράσουν δημιουργικά μακριά από τυφλές συντεχνίες οι οποίες τελικά το μόνο που θα κάνουν είναι να συσσωρεύουν την κουλτούρα σε συγκεκριμένο χώρο μόνο. Ε, και αυτό το τελευταίο αν συμβεί θα είναι δυστυχές και θα επιτείνει τη μετριότητα. Ε, πρέπει να κάνουμε το παν για να ε, έχει περισσότερος κόσμος πρόσβαση στη κουλτούρα, αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι όποιος έχει κάτι να πει, έχει μια αφήγηση, μια πρόταση καλλιτεχνική, να μπορεί να το κάνει σεβόμενη την έμπνευση, το ταλέντο και την ευφυΐα τους. Ε, εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε αυτές τις δράσεις. Ευχαριστώ για αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που είπατε και πιστεύω ότι πραγματικά αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση. Είναι θέμα πρόσβασης αλλά και ευκαιριών και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα ταλέντα, τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες και να σεβαστούμε και την ιδιαιτερότητα του καλλιτεχνικού κλάδου. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απαραίτητο και πολύ σημαντικό και ο πολιτισμός εκφράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν γίνεται ελεύθερα και με μια προσωπική έμπνευση και τη δυνατότητα να μην ε, ε, περιορίζεται αυτό σε καλούπια. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και τώρα ο κύριος Γύρι Σέστακ από την Γερουσία της Τσεχικής ε, Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Επιστημών Πολιτισμού, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αναφορών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η σημασία των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων ε, για την κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητη. Θα ήθελα όμως εδώ να ασχοληθώ ιδιαίτερα με ένα θέμα το οποίο μάλλον συνδέεται με τις κομμουνιστικές εμπειρίες πολλών κρατών και με τον ρόλο του παρελθόντος ε, στον πολιτισμό, διότι Η δική μας εμπειρία μας δείχνει ότι ο πολιτισμός συνδέεται με το βαθμό ε, ελευθερίας που έχει ένας λαός. Και βλέπουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας σε σχέση με τον πολιτισμό πολλά χρόνια μετά την πτώση του, στίχους, τείχους. Ε, και τα προβλήματα δεν ε, βρίσκονται μόνο στις ε, μεγάλες πόλεις. Τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν ε, και οι νέοι εδώ και χρόνια παρά το ότι η παλιά γενιά έχει πια πεθάνει. Υπάρχει το πρόβλημα της ε, ε, ρήμωσης των περιοχών της Υπέθρου. Οι νέοι πάνε στις μεγάλες πόλεις όπου έχουν ε, καλύτερες δυνατότητες να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους δυνατότητες. Αλλά έτσι χάνονται οι πολιτιστικές ρίζες. Κράτη που καταστράφηκαν ουσιαστικά από τη τα κομμουνιστικά καθεστώτα επί δεκαετίε έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού. Υπάρχουν περιοχές όπου έχει εκτοπιστεί ο αρχικός πληθυσμός που είχε όμως πολιτισμό αιώνων. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού ε, μιας χώρας. Έχουμε για παράδειγμα τον εκτοπισμό 3,5 εκατομμυρίων ε, Γερμανών, ε, γερμανόφωνων στην Τσεχία. Και μην ξεχνάμε ότι και οι εβραϊκές κοινότητες έχουν πάψει να υπάρχουν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό λοιπόν ε, έχει σημαδέψει ολόκληρες περιφέρειες ε, και οι ουλές υπάρχουν ακόμα. Μεταφέρθηκαν ε, λοιπόν πληθυσμοί σε άλλα μέρη της ίδιας χώρας ή σε άλλες χώρες με άλλες παραδόσεις που συχνά δεν έχουν καμία σχέση με τις παραδόσεις τις δικές τους. Υπάρχει πολύ λίγο ενδιαφέρον για τους δημόσιους χώρους στις περιπτώσεις αυτές και οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να παραμείνουν εκεί. Φαίνεται αυτό και στα ε, ρηπομένα κτίρια, τα εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και λοιπά. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με την πολιτιστική αυτή κληρονομιά. Υπάρχουν ακόμα μάρτυρες ε, εν ζωή. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα τραύματα. Περιοχές με πλούσιο πολιτισμό έγιναν ε, περιοχές ξεχασμένες από το χρόνο. Οι χώρες που δεν τα έχουν περάσει αυτά αδυνατούν να καταλάβουν την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Εδώ θέλουμε να συζητήσουμε κίνητρα, μέτρα και λύσεις για να στηρίξουμε τη συμμετοχή ε, των ανθρώπων στους δημιουργικούς τομείς. αλλά θεωρώ σημαντικό να αναφέρω το πρόβλημα αυτό, διότι είναι και αυτό θέμα που αφορά τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Πρόκειται και ευρωπαϊκό φαινόμενο, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και φυσικά πρέπει να προωθήσουμε και ένα μεγαλύτερο διάλογο δεν το λαμβάνουμε επαρκώς υπόψη, παρά το γεγονός ότι έχει σχέση και με άλλες πραγματικότητες και τελείως διαφορετική τοπική πραγματικότητα, νέα κέντρα και κυρίως ε, νέες γενιές. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο ε, πρέπει να το αναπτύξουμε και εν ώψη του πολιτιστικού, του έτσι πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο που είναι εξίσου πολύτιμο και αυτή είναι μεγάλη πρόκληση. Ωραία. Με αυτό νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με τους ομιλητές του πάνελ, αλλά Έχουμε τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Έχω δύο αιτήματα. Αν θέλει κάποιος άλλος να μου το πείτε τώρα, να δώσω λοιπόν το λόγο για δύο λεπτά στον καθένα. Στην κυρία Βίλστρομ καταρχάς, από τη Σουηδία, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ε, να σας ευχαριστήσω για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ε, και παρεμβάσεις. Έχω μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει πρόταση για ψηφιακό πλαίσιο, δηλαδή τυποποιημένες δομές για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εννοώ δηλαδή πώς μπορεί να γίνει πιο προσβάσιμη η ψηφιοποιημένη πολιτιστική κληρονομιά, πώς, ε, μπορεί, πώς μπορούμε να την ε, μοιράσουμε, να τη διαδώσουμε καλύτερα ή να χρησιμοποιηθεί ε, σε έρευνες. Η έλλειψη ενός τέτοιου πλαισίου μπορεί να οδηγήσει στο οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι να ψηφιοποιούν με διαφορετικό τρόπο την πολιτιστική κληρονομιά και να την κλειδώνουν, να μην είναι ανοιχτά προσβάσιμη. Μας ενδιαφέρει δηλαδή και στον τομέα αυτών η διαλειτουργικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν γίνονται ε, σχετικές εργασίες στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και μια απάντηση, να ακούσουμε και την άλλη παρέμβαση. Σουζάνα Μπαντέζοβαν λέω σωστά το όνομά σας, και από την Τσεχική Δημοκρατία, ε, από την Ομάδα των Φιλελευθέρων, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς εσάς κυρία Πρόεδρε για την ε, πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ σε αυτή τη συνεδρίαση. Θέλω να ευχαριστήσω και την Τερέζα από το, τη γραμματεία της Τσεχικής Γερουσίας που μας συνοδεύει και μας ε, διοργάνωσε όλη αυτή την αποστολή. Δύο είναι οι βασικές σκέψεις που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και τις θεωρώ σημαντικές. Πρώτον, κάτι που είναι κάπως διαφορετικό, αλλά αξίζει ωστόσο να αναφερθεί πιστεύω και αναφέρομαι στην κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων των μεταναστών. 78% το των παιδιών στα κέντρα προσφύγων είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ας διασφαλίσουμε ότι αυτά τα παιδιά θα καταχωριστούν, θα ταυτοποιηθούν, δεν θα χωριστούν από τους γονείς τους αυτοί που τους έχουν, ότι δεν θα χαθούν και δεν θα γίνουν θύματα ε, κακοποίησης. Ζητώ συγγνώμη, αλλά προσπαθώ να αξιοποιήσω αυτή την πλατφόρμα και αυτό το βήμα διαλόγου που μου δίνεται για να σκεφτούμε όλοι για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω έχει να κάνει με κάτι που είπε και η κυρία Κώστα, ότι πρέπει δηλαδή να χτίζουμε γέφυρες και να μην τις γκρεμίζουμε με πολέμους. Συμφωνώ απολύτως. Ο πολιτισμός είναι αυτός που ενώνει τους ανθρώπους, η μουσική ε, ξεπερνά τα σύνορα, η τσεχική δημοκρατία έχει πάρα πολλά να προσφέρει, έχουμε εξαιρετικούς ε, μουσικούς ε, συνθέτες, πασίγνωστους όπως και άλλα ευρωπαϊκά έθνη άλλωστε, θυμάμαι ως παιδί ότι έβλεπα την Eurovision, τη Eurovision στην τηλεόραση. Και τότε βλέπαμε το καλύτερο, ε, τον ανθό τον της μουσικής παραγωγής των ευρωπαϊκών ε, κρατών, ε, σε μια προσπάθεια να μοιραστούμε τις αξίες μας. Νομίζω ότι το να παρίσταται κανείς σε μια καλή συναυλία, αυτό είναι κάτι που ενθαρρύνει την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε τη, τη φιλία, την αγάπη, την ε, κουλτούρα, τον πολιτισμό. Εάν βρίσκονται χρήματα για όπλα, ε, τότε μπορούν να βρεθούν και για διεθνείς συναυλίες. Και αυτό προτείνω ως συνεισφορά να διοργανωθεί το Ευρωπαϊκό Έτος ε, Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Νομίζω ότι μια τέτοια διεθνή συναυλία θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία αυτή η φράση. Αφού υπάρχουν χρήματα για όπλα, πρέπει να υπάρχουν και χρήματα για τον πολιτισμό. Πολύ ωραίο μήνυμα. Η συνάδελφος αντιπρόεδρος ε, από το ΕΛ και η κυρία Σβεντρόβα από την Σλοβακική Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι τρεις ε, εκπρόσωποι της Τσεχίας παίρνουν το λόγο ένας μετά τον ε, άλλο και χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Η κουλτούρα, ο πολιτισμός είναι κάτι που μας ενώνει. Ένα άλλο στοιχείο που μας ενώνει είναι το γεγονός ότι σε κάθε χώρα, αλλά και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να αγωνιστούμε για οικονομικούς πόρους. Αυτή η Επιτροπή, υπό την Προεδρία τη δική σας κυρία Κώστα, ανέκαθεν έδινε αυτόν τον αγώνα εξέβρεσης πόρων για την προστασία και στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των νέων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών σχεδίων. Έχουμε 10 χρόνια πλέον το κινηματογραφικό βραβείο Lux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ανταμείβει την ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία. Είναι, ένα, είναι καλή ιδέα η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια για να στηρίξουμε τον ασιατικό κινηματογράφο. Θα συνεργαστούμε και για το έτος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και η ιδέα αυτής της κοινή συναυλίας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Καταρτίζουμε τα διάφορα προγράμματα, τα διάφορα έργα και είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί ένα τέτοιο project. Ε, ε σας ευχαριστώ γιατί αναφερθήκατε και στην ε, ψηφιοποίηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Είναι κάτι το οποίο συζητούμε στην τσεχική δημοκρατία. Η ψηφιοποίηση ε, συνδέεται με τη διατήρηση της ποιότητας της αρχικής εργασίας. Άλλωστε, σε ό,τι αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους και πιο συγκεκριμένα στον ε, καταβλισμό του Καλέ ε, στους οποίους αναφερθήκατε, πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, είμαστε μέλη της διακλαδικής ομάδας για τα παιδιά των προσφύγων και ασχολούμαστε με τη βοήθεια και στήριξη όλων αυτών των παιδιών. Μιλούμε συνεχώς ε, για αυτό το πρόβλημα και διαδίδουμε πληροφορίες. Σας ευχαριστώ που το αναφέρατε και προσδοκώ μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ κυρία Σφεντρόβα και γιατί υπενθυμίσατε αυτή την κοινή δέσμευση για τους ανήλικους. Υπενθυμίσατε ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η ε, ανήλικοι είναι ένα θέμα που απασχολούν ε, όλους μας αυτή τη στιγμή και ε, φυσικά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχουμε και αυτή λοιπόν την ε, ομάδα για τους ανήλικους που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, περιλαμβάνει συναδέλφους ε, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά με κάρσιο τρόπο και προσπαθούν να δώσουν μια νέα όθηση και να συμπεριλάβουν το θέμα των ε, ανηλίκων σε όλες τις επιτροπές. Το λέω γιατί συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε μέχρι πριν από λίγο η κυρία Σβεντρόβα. Ο κύριος Μπλός έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Δεν είχα σκοπό να παρεύω για δεύτερη φορά, ωστόσο καλούμε να το κάνω μετά την παρέμβαση του Τσέχου ε, συναδέλφου της ε, και στη συνέχεια ε, το τόνισε αυτό και συνάδελφος του Intergroup. Δεν βλέπω πώς μπορεί να κατηγορηθεί η Γαλλία ε, για την πολιτική της. Εγώ είμαι ερετός στο Παρίσι ε, και γνωρίζω ότι η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχει αυξήσει και πάρα πολύ μάλιστα σημαντικά ε, τα επιδόματα για την παιδική ηλικία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε όλους τους νομούς της Γαλλίας, έτσι ώστε να στηρίξει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των ε, παιδιών αυτών. Από εκεί και πέρα, ε, γι' αυτό παίρνω το λόγο, γιατί δεν καταλαβαίνω καθόλου ε, πώς θα μπορούσε κανείς να κατηγορήσει τη Γαλλία και πού θα πώς θα μπορούσε να ευσταθεί ένα τέτοιο επιχείρημα με δεδομένη ε, την αύξηση του προπολογισμού ε, της Γαλλίας για τέτοιου είδους ενίσχυση και τέτοιου είδους επιδόματα. Ευχαριστώ πολύ μπορώ να δώσω και το, λόγο στην κυρία Σπετρόβα, αλλά νομίζω ότι το, το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι ένα πρόβλημα που έχουμε σε πολλέ χώρε. Είναι ένα θέμα που αφορά χιλιάδε παιδιά και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο από εμά ο οποίο είναι χωρί ευθύνε. Ο αναμάρτητος πρώτο στο Λιθοβαλέτο. Υπάρχουν ευθύνε για όλου μα. Το λέω για την Ιταλία που ε, 150.000 πρόσφυγε. Υπάρχει πρόβλημα. Ε, παρά το γεγονό ότι η Ιταλική αλληλεγγύη, επιτρέψτε μου αυτό το μικρό σοβινισμό, είναι κάτι που δεν επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ξέρω λοιπόν ότι υπάρχει το πρόβλημα, δεν ήταν κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, καλό είναι να το αναφέρουμε και φυσικά μα ανησυχούν όλου ότι υπάρχουν κάποια ε, καταστάσεις ε, πολύ ε, σημαντικές στην Ευρώπη και ξέρουμε ότι είναι ένα φλέγον ζήτημα το θέμα των ανηλίκων. Δεν ήταν συγκεκριμένη κατηγορία νομίζω, απλώς ήταν μια διαπίστωση για καταστάσεις που υπάρχουν και σε άλλα σύνορα. Παρακαλώ. Oh, oui, merci. Je Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, θέλω να απαντήσω. Δεν κατηγόρησα τη Γαλλία ότι κάνει κάτι εσφαλμένο ή λάθος. Αντιθέτως, λέμε ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σας βοηθήσουμε, να φροντίσετε, να φροντίσουμε όλοι τους ανηλίκους και κυρίως τους ασυνόδευτους και να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε ε, ε, αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Νομίζω ότι πρόκειται περί παρανόηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βλός. Ναι, ναι, δεν απαντούσα σε εσά, κυρία μου. Απαντούσα στο μέλος του ε, της ε, Τσεχικής Βουλής. Δεν κατάλαβα την παρέμβαση ε, του Τσέχου συναδέλφου σας διαβεβαιώ και σας καθησυχάζω κυρία μου ότι τα λόγια μου δεν, στρέφονται δεν στρέφονταν εναντίον σας. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει λόγος τώρα να ανοίξουμε συζήτηση. Έχουμε ευκαιρίες να το συζητήσουμε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω με κάτι που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το οποίο είμαι ιδιαίτερα περηφανή, διότι η πρωτοβουλία ξεκινά από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εγκρίναμε δύο πολύ σημαντικά ψηφίσματα ε, που ε, αφορούν τους ε, ανήλικους πρόσφυγες. Το πρώτο ψήφισμα προέκυψε βάση του εξή τυχαίου. Σήμερα μόνο το 2% της ανθρωπιστικής βοήθειας, δηλαδή αναφέρομαι και σε πρόσφυγες που βρίσκονται εκτός Ευρώπης, ε, πηγαίνει στην πρόσβαση στην παιδεία αυτών των παιδιών. Υπάρχουν ε, ε, χιλιάδες παιδιών που βρίσκονται σε στρατόπεδα προσφύγων σε πονίδιστες συνθήκες και ορισμένες φορές ε, πολλοί από αυτούς φιλοξενούνται στις φτωχότερες ε, χώρες ε, στο Λίβανο, στην Ιορδανία και τα γνωρίζουμε. Αυτό δεν τιμά την Ευρώπη και το λέω ως Ευρωπαία, ούτε ως Ιταλίδα, ούτε ως οτιδήποτε άλλο. Και εμείς ε, λοιπόν γκρίναμε ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα με την Επιτροπή Ανάπτυξης και ε, λάβαμε 153 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ από αυτή την εκστρατεία που ξεκινήσαμε που λεγόταν έντουκα ε, ε, και προτείναμε 4-4-4 να έχουμε δηλαδή τουλάχιστον 4% δεν είναι ε, αρκετό αλλά τουλάχιστον ως πρώτη χώρα περιοχή δωρητής ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε κάτι παραπάνω ε, για να αποφύγουμε και τη ριζοσπαστικοποίηση, τις σειράξεις, ε, να ε, υπάρχει πρόληψη μέσω της παιδείας. Η άλλη δρέση που προωθήσαμε και αυτή πάλι μέσω ψηφίσματο που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιε χώρε ήταν ιδιαίτερα δραστήριε και μάλιστα θα ήθελα εσεί ω εθνικοί βουλευτέ να πιέσετε και τι κυβερνήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, είναι ένα ψήφισμα που λέγεται εκπαιδευτική διάδρομη ε, για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, για μια χαμένη γενιά των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αυτέ τι δυσκολίε. Ζητήσαμε από τα ε, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, απάντησαν αρκετά πανεπιστήμια, όχι όλα και όχι πολλά, αλλά έχουμε ένα πρώτο αριθμό. Και το UNIMED, το Πανεπιστήμιο της Μεθοσογείου δέχτηκε να φιλοξενήσουν αυτούς τους φοιτητές, κινδυνεύουν να μην καταφέρουν να σπουδάσουν, γιατί εδώ και δύο-τρία χρόνια αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Μαζί με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες, μαζί ε, με την ε, διάσκεψη των διευθυντών σε εθνικό επίπεδο, μαζί με ανθρωπιστικές οργανώσεις, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και νομίζω ότι πρέπει σήμερα να αποστείλουμε αυτά στις ε, ενδείξει, αυτά τα σήματα στους ανθρώπους αυτούς που ζουν στα παράλια της Μεσογείου, που βλέπουν την Ευρώπη ως ένα κλειστό φρούριο που κλείνει όλο ένα και περισσότερο. Είμαστε περήφανοι λοιπόν για αυτά τα ψηφίσματα. Να δούμε τώρα από εκεί και πέρα πώς μπορούμε να εξετάσουμε κάποιες καταστάσεις. Σίγουρα όμως μας ανησυχεί το γεγονός ότι οι ανήλικες συχνά, όπως κατήγγειλε η UNICEF και άλλες διεθνείς οργανώσεις, δεν προστατεύονται παρκώς και δεν γίνονται σεβαστές διεθνείς συμβάσεις που έχουμε υπογράψει όλοι. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο ε, έχουμε αναλάβει. Η Julie Ward ήθελε το λόγο και σιγά σιγά θα περάσουμε στα συμπεράσματα. Να αναφερθώ σε αυτό το θέμα το των ασυνόδευτων ανηλίκων και να μιλήσω συγκεκριμένα για αυτό που συμβαίνει στο Καλέ και στη Δουνκέρκη, διότι έχω επισκεφτεί τα μέρη αυτά τρεις φορές και Πιστεύω ότι ο πολιτισμός έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μας με ανθρώπους που δεν έχουν τα δικά μας πλεονεκτήματα. Είτε μιλάμε για άστεγους στις πόλεις μας, είτε μιλάμε για πρόσφυγες ε, που βρίσκονται στο τέλος μιας μακράς διαδρομής. Είμαι περήφανη για τη δουλειά που κάνουμε εδώ. Πρέπει να πω όμως ότι ως Ευρωβουλευτής ε, του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είμαι περήφανη για τη χώρα μου. Δεν είμαι περήφανη που οι κυβερνήσεις μας δεν μοιράζονται ίσα το βάρος και σε κάποιε περιπτώσεις δεν κάνουν όσα μπορούν να κάνουν. Έχοντας επισκεφτεί το Κάλε και τη Δουνκέρκη, μου έκαναν εντύπωση οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι εθελοντέ, οι δάσκαλοι που ε, στον ελεύθερο τους χρόνο στις αργίες τους ε, διδάσκουν ε, διάφορα μαθήματα, όχι μόνο αγγλικά και γαλλικά, αλλά και ε, χορό, μαθηματικά, επιστήμες, γεωγραφία. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους αναλαμβάνουν εκεί που οι κυβερνήσεις έχουν αποτύχει. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε μια πλατφόρμα στους ανθρώπους αυτούς, ε, να ακούσουμε τις ιστορίες τους και ε, να τους δώσουμε αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αποτύχαμε. Αποτύχαμε εμεί ε, και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν αναλάβει και πολλέ από αυτέ τι μη κυβερνητικέ οργανώσει χρησιμοποιούν τον πολιτισμό και τι τέχνε διότι είναι κάτι που βοηθάει να εξανθρωπίσει ανθρώπους που έχουν χάσει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Έχουμε κρίση αλληλεγγύης, ε, ε, όχι κρίση προσφυγική. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές αυτό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βαραίνει τη συνείδησή μας ε, και τα θεσμικά όργανα όμως και τις πολιτικές ομάδες, ε, βαραίνει όλη την Ευρώπη. Είναι ένα γενικό ζήτημα το οποίο δεν θα πρέπει να αφήσουμε να ε, ε, χαθεί στη λύθη. Πρέπει να μην σιωπήσουμε, να πούμε σαφέστατα πώς έχουν τα πράγματα και να έχουμε και τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και τις ανεπάρκειες της Ευρώπης. Σήμερα βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός είναι ε, πολύ πολύτιμα αγαθά και πρέπει ε, να προσπαθήσουμε να τα διατηρήσουμε εάν πραγματικά θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε κάτι λογικό στις επόμενες γενιές. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Σας ευχαριστώ ε, εκ βάθους καρδίας για τη συμμετοχή. Ε, θα ήθελα να σταθώ σε κάποια πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα πω όλα ή αν υπάρχει κάποιο συνάδελφος ο οποίος θα ήθελε να απαντήσει. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μόργανο ή κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Βλέπω ότι δεν θέλει κανείς. Εγώ δεν διανοούμε καν να πω ότι ολοκληρώνεται τη συζήτηση. Θα προσπαθήσω απλώς να δω κάποιες προτάσεις και να απαντήσω ίσως και σε ε, μία ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω, διότι με ε, άγγιξαν κάποιες παρεμβάσεις και τις θεωρώ πολύτιμες. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να προδώσουμε τον πολιτισμό ως αγαθό αυτό καθεαυτό. Να θεωρείται αγαθό αυτό καθεαυτό και όχι ως αγαθό το οποίο έχετε να συμπληρώσει άλλους τομείς. Συμφωνούμε να μιλάμε για τον πολιτισμό, αλλά για τον πολιτισμό στην οικονομία, στην τεχνολογία κλπ. Ο πολιτισμός είναι ένα αγαθό αυτάρκες, αυτούσιο και πρέπει λοιπόν να έχουμε κάτι το οποίο θα σέβεται την ελευθερία των πολιτιστικών δικαιωμάτων, τα οποία παρεπιπτόντως περιλαμβάνονται και στα θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα ε, ε, της ελεύθερης έκφρασης ε, μέσω δημιουργικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργεί και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Και αυτό είναι το πρώτο μας καθήκον. Δεύτερον, να υπάρχει μια δημοκρατική αντίληψη του πολιτισμού. Δηλαδή να υπάρχει όλο και όσο το δυνατόν περισσότερη δυνατότητα πρόσβασης. Και όπω είπαν και οι εμπειρογνώμονες, δεν σημαίνει η πρόσβαση ότι είμαστε απλώ θεατέ. Σημαίνει ότι συμμετέχουμε και εμείς. Το audience development ε, στην αρχή ήταν audience building. Εμείς το κάναμε development γιατί αυτό μας επιτρέπει να έχουμε διάφορε διαστάσει. Η διεύρυνση του κοινού βεβαίω η δυνατότητα να αναπτύξουμε τον πολιτισμό ε, του κοινού. Υπάρχει θέμα επιμόρφωσης και κατάρτισης των παιδιών. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί υπήρχε και μια έκκληση να είμαστε δημιουργικοί. Εγώ έχω δει από κοντά εμπειρίες στην Ιταλία, στη Σουηδία, υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο παιδιών που από πολύ μικρά εκπαιδεύονται και μαθαίνουν για παράδειγμα να παρακολουθούν ε, όπερα και από, από τριών χρονών και πάνω που σημαίνει ότι υπάρχει ένα νέο κοινό ε, μορφωμένο και κατά την άποψή μου, για παράδειγμα, στα σχολεία θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να μαθαίνουν να παίζουν ένα μουσικό όργανο τα παιδιά. Ε, όλες αυτές οι ευκαιρίες, όλες αυτές οι δεξιότητες ε, ε, που πολύ συχνά λέει η Τζούλη, δημιουργικές δεξιότητες, είναι ε, ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη ζωή, για να είμαστε ε, πλήρεις πολίτες και να νιώθουμε πάντα ότι είμαστε ενεργοί πολίτες. Μου αρέσει όμως και το θέμα του audience engagement, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι να έχουμε ενεργό συμμετοχή, η οποία με τη σειρά της θα δημιουργήσει και άλλα πράγματα. Τρίτον, η διάσταση του πολιτισμού ως πολιτιστική βιομηχανία, ως οπτικοακιστική βιομηχανία, παραγωγική βιομηχανία και ε, η δύσκολη αντιπαράθεση με την ε, ψηφιακή πρόκληση είναι το άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ε, δράσης μας. Ενώ παραδοσιακά στο παρελθόν αυτό περιοριζόταν στην οπτικοακουστική βιομηχανία. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπαν αρκετοί από εσά, έχουμε και την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία. Έτσι διευρύνθηκε το φάσμα, διότι υπάρχει μια ενδιάμεση περιοχή δημιουργικότητας νέων υπηρεσιών, ακόμα και σε άλλου τομεί ε, καινοτομία ε, μέσω ψηφιακών ε, δομών κλπ που έχουν όμως ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα και μπορούν να είναι οικονομικής φορείς αλλά και φορείς ε, κοινωνικής καινοτομίας και κοινο, ε, ε, η οποία θα διαχέεται και σε άλλους τομείς όπως είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει το θέμα της κατάρτισης και των δεξιοτήτων. Ίσως να είπαμε ελάχιστα και αυτό δεν υπάρχει μόνο θέμα παιδείας, να μάθουν τα παιδιά την τέχνη κλπ. Αλλά υπάρχει και η αξιολόγηση ε, όλων αυτών των εξαιρετικών δεξιοτήτων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ε, εστιατόρες, ε, εμπειρογνώμονες, ε, διαχειριστές πολιτιστικών αγαθών. Προηγουμένως είπαμε ότι τα μουσεία, η γκαλερί τέχνης δεν πρέπει να είναι πια αυτά που είναι σε κάποιες χώρες, ε, παραδείγματος χάρη στη δική μου που ήταν λίγο πιο συντηρητικό στα πολιτιστικά αγαθά, αυτή τη στιγμή έχει μια τεράστια όθηση προς την άλλη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, εγώ γνωρίζω υπάρχουν αυτά τα σημαντικά δίκτυα, το e το δίκτυο των μουσείων. Πλέον υπάρχουν νέοι διευθυντές μουσείων οι οποίοι έχουν πολύ καλές ε, ε ικανότητες, ε, πολύ ισχυρέ ικανότητες. Ε, είναι ικανότητες λοιπόν τις οποίες πρέπει να προωθήσουμε και να τους εκπαιδεύσουμε. Υπάρχει μεγάλη πρόκληση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είπε, ίσως ο εμπειρογνώμονας από τη Βαλονία. Διαχείριση στη συμπαραγωγή. Υπάρχουν δηλαδή νέα επαγγέλματα ε, που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Κάποια τα είδα και στις πολιτιστικές πρωτεύουσες, διότι στην αρχή οι πολιτιστικές πρωτεύουσες ήταν απλώς ε, κάποιες εκδηλώσεις της πόλης ε, σε μια χρονιά. Στην πραγματικότητα, στο τέλος έγιναν κάποιες ολοκληρωμένες ομάδες, οι οποίες πλέον έχουν και δίκτυο, που μπόρεσαν να βοηθήσουν τις πόλεις μέσω μιας διαφορετικής ανάγνωσης σε πολιτιστικό επίπεδο των δυνατοτήτων μιας πόλης και σε θέματα ε, υπήρξαν πόλεις οι οποίες κατάφεραν να σκεφτούν, για παράδειγμα, τη νέα του εκβιομηχάνισμα. Ε, το Λίβερπουλ, η Γλασκόβη, ε, η Ρουρ. Ε, πρόκειται για πόλεις οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία και αυτή τη στιγμή προωθούν έργα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, χάρη αν μου επιτρέπετε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν στο εσωτερικό τους και τη δυνατότητα να, να χρηματοδοτήσουν και να υποστηρίξουν και παρεμβάσεις για την πολιτιστική κληρονομιά, για νεοφυείς επιχειρήσεις, για επιτροπές επιτόπου, για πολιτιστικό περιεχόμενο. Ξέρουμε βεβαίως ότι στα διαρθρωτικά ταμεία υπάρχουν δύο ή τρεις γραμμές προπολογισμού που προβλέπουν και τα θέματα αυτά και τη δημιουργική βιομηχανία. Πολλές περιοχές στην Ευρώπη, πολλές περιφέρειες ε, ε, εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα κονδύλια για lab, για κόμβους, ε, για τσεκ, για νέους, για υποτροφίες εργασίας κλπ. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές δυνατότητες. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ένα ανώτατο όριο 5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις για τον πολιτισμό και δεν είναι μόνο διαδικασίες αναστήλωσης, αλλά να έχουμε κάποιες άλλες δυνατότητες σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο διαχείρισης. Λοιπόν, πολιτιστική κληρονομιά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν ήδη στην Ευρώπη και είναι εξαιρετικά. Ορισμένε φορέ δεν διασταυρώνονται αρκετά. Και κάποιε από τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να. Ε, οι εθνικοί Ευρωπαϊκοποιήσουμε τα ε, πολιτιστικά ιδρύματα για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένε φορέ μένουν πολύ στο περιθώριο και δεν μπορούν να ε, αξιοποιήσουν τι ανταλλαγέ. Παραδείγματο χάρη, εγώ ανακάλυψα πρόσφατα και το γνωρίζατε το δίκτυο Excite. Θα μου πείτε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και γνωστό. Εγώ το ανακάλυψα πριν από δύο χρόνια. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με το ακρόνιμο Excite ε, μουσείων επιστήμης. Στην πραγματικότητα δεν είναι μουσεία επιστήμης, είναι χώροι στους οποίους εκπαιδεύουμε στην επιστήμη. Σιγά σιγά ε, να έγιναν 90, ε, είναι εξαιρετική η καινοτομία στις εκπαιδευτικές μεθόδους και έχουν γίνει και fab lab αυτή τη στιγμή. Πρόκειται λοιπόν για κινήματα τα οποία υπάρχουν και αυτό προσπαθώ να σας πω με αυτό το παράδειγμα. Παράδειγμα για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο λέγεται Πώ το λένε τώρα, το ξέχασαμε, πώς το ξέρετε εσεί για την πολιτιστική κληρονομιά. Τέλο, πάντων θα μου ήρθει. Ε, υπάρχουν λοιπόν δίκτυα όχι, όχι αυτό. Για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ε, το οποίο μεταξύ άλλων ασχολείται και με digital humanities, ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές. Ε, πρόκειται για κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται για ερευνητικά ιδρύματα ή, ε, ή άλλης δεν είναι μόνο ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή, τα οποία έχουν ε, αφιερώσει πάρα πολλούς πόρους από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Αυτό σημαίνει ότι σε διεθνές επίπεδο μπορούν να μοιράζονται ε, μια μεγάλη δέσμευση για την ψηφιοποίηση της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Απαντάω στη Σουηδή συνάδελφο που έθεσε το ερώτημα αυτό. Είναι σε πολλούς τομείς. Στην έρευνα, στον Ορίζοντα 2020 υπάρχουν πόροι, υπάρχουν πόροι στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα και στην Εθνική ε, στο Εθνικό Ψηφιακό Θεματολόγιο που χρηματοδοτούν και σε άλλα. Και υπάρχει και το πρόγραμμα Ευρωπαϊνα, στο οποίο η Γενική Διεύθυνση Connect ε, τροποποίησε ε, την λεγόμενη υπηρεσία Ευρωπαϊάνα, στην πούμε υπηρεσία, και προβλέπεται η συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών χωρών και υπάρχουν και κάποιες επιλογές όσον αφορά την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού, της πολιτιστικής κληρονομιάς που θέλουν να είναι ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα εμβαθύνετε αυτά και επίσης υπάρχει και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, Κινηματογραφικών Εθουσών, Μουσείων και έγινε ένα αφιέρωμα μαζί με την Ευρωπαϊάνα για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, στο οποίο όλες οι ε, κινηματογραφικές λέσχες διηγήθηκαν την ίδια ιστορία από τη δική τους κοπιά. Τι σημαίνει αυτό και έρχομαι και σε κάτι άλλο ε, το οποίο ε, αφορά το πρόγραμμα το οποίο τροποποιήθηκε λίγο από τον Επίτροπο Ναβράτσετς και άνοιξε και στους νέους αυτή η λεγόμενη περιβόητη νέα αφήγηση για την Ευρώπη, το New Narrative for Europe. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να διηγηθούμε λίγο καλύτερα για να γίνει γνωστό και να υπάρχει και κατάλληλη συμμετοχή και από τους νέους ε, ένας νέος τρόπος να ε, αφηγούμαστε την Ευρώπη. Ίσως θα έπρεπε να σταματήσω εδώ. Πιστεύω ότι όπως ε, θα είδατε προσπαθήσαμε να μοιραστούμε μια στρατηγική, η οποία αυτή τη στιγμή έχει αυτούς τους τέσσερις βασικούς ε, άξονες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, αλλά δεν εξαντλείται εκεί. Κυρίω μα ενδιαφέρει βέβαια ε, η οικονομία, αλλά δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα και παίξαμε λίγο και το παιχνίδι να το κάνουμε αυτό μαζί με την Επιτροπή Βιομηχανία. Κάποιοι είχαν και κάποιε αμφιβολίε, αλλά για μένα ε, προέκυψε το εξή. Τελικά, η ε, βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να ασχοληθεί και με την πολιτιστική βιομηχανία. Όχι να πάρουμε τα λίγα χρήματα που έχει η Δημιουργική Ευρώπη. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι ε, ξεκίνησε επισήμως και λογικά σε λίγο θα ξεκινήσουμε και θα καθοριστεί και η πορεία. Η πρώτη προκήρυξη για τον διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για το νέο μέσο για την εγγύηση για την Ευρώπη για τα εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία θα δανειοδοτήσουν τον τομέα ε, της δημιουργικής ε, και πολιτιστικής βιομηχανίας. Είναι κάτι το οποίο προβλεπόταν στη δημιουργική βιομηχα... Ε, Ευρώπη. Ελπίζω να υπάρχει και κατάλληλη γεωγραφική κατανομή και να περιληφθούν όλοι οι κλάδοι και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και εκεί θα δούμε πώς αυτός ε, ο κόσμος ε, των ε, τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών, χρηματοπιστωτικών ιδεμάτων θα ανταποκριθεί. Η προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού συνοδεύεται και από μία άλλη δράση ικανοτήτων αυτών των ε, ιδρυμάτων. Υπάρχει λοιπόν εμπειρογνωμοσύνη η οποία θα ε, συνοδεύσει αυτή την προσπάθεια γιατί ξέρουμε ότι αυτό δεν υπάρχει στην πραγματικότητα χωρίς αυτό. Ε, τελευταίο στοιχείο η πολιτιστική διπλωματία. Είναι άλλος τομέας αυτός, το λέω γιατί θα μπορούσαμε ίσως αυτές τις στρατηγικές να τις έχουμε και σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρώπη ε, στοιχηματίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική ασφάλεια, σε εξωτερική πολιτική, πολιτική και πολιτική της ολοκλήρωσης και της μετανάστευση, εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη σε όλες τις ε, σχέσει, τι εταιρικέ σχέσεις μεταξύ Ευρώπη και του υπόλοιπου κόσμου ε, ο άξονας, του άξονα συγγνώμη, του πολιτισμού, της παιδεία, ε, και ε, τα ψηφιακά ζητήματα φυσικά είναι το μεγάλο ερωτηματικό για το οποίο αναρωτιόμαστε όλοι. Πολλοί το θέσατε αυτό το θέμα. Εμεί αυτή τη στιγμή συζητούμε την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ε, εκτιμούμε το γεγονό ότι γίνεται προσπάθεια από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την πρότασή μα. και εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε κάποια αγαθά να προστατεύονται, σίγουρα να προστατεύονται οι νέοι αλλά και οι, δημιουργοι... οι συγγνώμη, αλλά η δημιουργικότητα και άλλα και γιατί οι πλατφόρμες, κυρίως οι πιο προηγμένες και αυτοί οι οποίοι παράγουν περιεχόμενο και ε, στην πραγματικότητα συμμετέχουν κιόλα, ε, το έθεσε και προηγουμένω η Χέλγα Τρούπελ, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε ε, στις πλατφόρμες ε, που μοιράζονται περιεχόμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, τα VOD όμως περιλαμβάνονται, που σημαίνει ότι πρέπει να σέβονται το εξή. Κανόνες, προστασία των ανηλίκων, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, κάποια θέματα που αφορούν τη διαφήμιση και το πιο ενδιαφέρον, για πρώτη φορά λέγεται κάτι που περίμεναν πολλές χώρες. Σίγουρα η Γαλλία, η Γερμανία κλπ. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν από αυτούς τους κυρίους πόρους ε, που θα επενδύσουν και πάλι στον πολιτισμό. Διότι νομίζω ότι έτσι πρέπει από πλευράς πολιτικής αξιοπρέπειας να γίνει. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι όλα αυτά είναι εν εξελίξη. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, κάτι μου λένε εδώ. Μισό λεπτό να δω τι είναι. Ναι, βεβαίως υπάρχει και αυτό. Εγώ πιστεύω για άλλη μια φορά ότι αυτή η άμεση διάλογη είναι μια ε, ε, πρώτη ευκαιρία. Δεν είναι η τελευταία φορά που θα συναντηθούμε. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Το ξέρετε το δρόμο για τις Βρυξέλλες καλά. Είναι μια πρώτη συνάντηση. Ελπίζω να έχουμε και ακροάσεις και στις δικές σας επιτροπές πολιτισμού, στα κοινοβούλια σας, διότι σίγουρα βοηθά ε, αυτό, μια ανταλλαγή απόψεων που πολλές φορές είναι πολύ περιορισμένη. Πιστεύω ότι εμείς πρέπει καλύτερα να υλοποιήσουμε το σύστημα, ε, τη φάση ε, εκ των άνω προς τα κάτω των αποφάσεων και όχι μόνο, μάλλον από κάτω προς τα πάνω και όχι μόνο εκ των άνω προς τα κάτω και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο και κυρίως τη Γενική Διεύθυνση των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια που ε, εκπροσωπούνται εδώ στο ύπατο επίπεδο, διότι χωρί αυτού δεν θα μπορούσαμε να είχαμε διοργανώσει όλα αυτά τα πράγματα. Και την υπομονή με την οποία διοργάνωσαν όλα αυτά τα πράγματα και μα υποστήριξαν, όπω επίση και τι ικανότητε του. Είμαι ευγνώμων λοιπόν, μπορούμε να είμαστε πιο δημιουργικοί στι σχέσει μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμεί είμαστε στη διάθεσή σα. Σα ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσία σας εδώ και για την πολύ μεγάλη συνεισφορά σας. Θα σας ε, διανύμουμε έγγραφα. Έχετε ήδη στο φάκελό σας τεκμηρίωση. Θα είδατε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά βεβαίως αν υπάρχουν κάποιες ε, ανάγκες για περαιτέρω τεκμηρίωση μπορείτε να μας τα ζητήσετε και να γίνει συνήθεια πια αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών κάποιοι νόμοι που μας ανακοινώσετε για τις χώρες σας να μας τους στείλετε, είναι πολύ σημαντική, ε, διότι νομίζω ότι αυτό βοηθά και την προοπτική μιας ευρωπαϊκής ε, πολιτιστικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ στο επανειδή.